Um, Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε και ας αρχίσουμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι τα ειδικά θέματα τα οποία θα ξεκινήσουμε. Um, το πρώτο επομένως στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση αυτής. Και σας ενημερώνω ότι θα μεταδίδεται στο ίντερνετ η συνδυασή μας εκτός από το κομμάτι που είναι και κλεισμένο. Και το χρονοδιάγραμμα που βλέπετε γραμμένο είναι ενδεικτικό χαρακτήρα και τα πράγματα θα είναι ρευστά, μπορεί να αλλάξουν. Και έχουμε σε εξή αλλαγέ στην διάταξη. Τα 5, 13 και 14 θέματα ε, δεν θα ζητηθούν, να αναβάλει τη ζητηθή του, ε, αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Οπότε θεωρώ που δεν υπάρχει ένσταση ότι εγκρίνεται η διάταξη Πολύ ωραία. Το επόμενο τώρα είναι οι ανακοινώσει σε σχέση με τη συνεδρίαση των συντονιστών σήμερα το πρωί, οι οποίοι απεφάσισαν. Σήμερα, με, βάση του κανόνε που έχει θέσει η διάσκεψη των Προέδρων στην απόφαση τη 5η ε, Μαρτίου 1998, αποφάσισαν για τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ειδικευμένων Φορέων και ε, προτείνουν στην Επιτροπή Τζούρι για να αποφασίσει τα ονόματα των υποψηφίων για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Επιτροπής προπολογισμών. Η ψηφοφορία γι' αυτό θα γίνει στη σημερινή μα συνεδρίαση. Επίση, συμφώνησαν να προσκαλέσουμε το Ελεκτικό Συνέδριο και τον Επίτροπο για τη Δίκηση και τον Προπολογισμό όταν επιβεβαιωθεί το ε, Σώμα των ε, Επιτρόπων να μα παρουσιάσουν ε, τα πορίσματα τη ειδική έκθεση του ελεκτικου συνεδριου Συνεδρίου 15-2019 για την εφαρμογή του πακέτου για τη μεταρρύθμιση του προσωπικού του 2014. Επίση, οι συντονιστέ ε, συμφώνησαν να συντάξουν μια γνωμοδότηση ω επιστολή για την Επιτροπή Αναφορών όσον αφορά την ε, αναφορά 0193 κάθε 2019 από τον Τζάμισον Γιάνγκ που είναι τσέχο, για του όρου που χρησιμοποιούν οι μη εμπορικοί φορεί συλλογή ε, πνευματικών δικαιωμάτων και μια γνωμοδότηση με μορφή επιστολή προ την Επιτροπή ΑΦΚΟ για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τη συμφωνία για την αποχώρηση. Ο πρόεδρος ή πρόεδρος θα είναι η προεδρος θα ειναι η για τα δύο οι συντονιστέ συμφώνησαν να ορίσουν τον κύριο Φράνκο Ρομπέρτη, σοσιαλιστή, ω ε, εισηγητή για την πρόταση ε, υποβολή στα κράτη-μέλη εγγράφων δικαστικών και εξοδικαστικών για αστικά και εμπορικά θέματα από την προηγούμενη θητεία. Επίση, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε τον συντονιστή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των παιδιών, την κυρία Εύα, την συντονιστή, λοιπόν, κυρία Εύα Κοπάτ, σε μια τη επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή μα, ενδεχομένω 27-28 Ιανουαρίου 2020. Επίσης, οι συντονιστές ανέκριναν το πρόγραμμα έρευνας της Τζούρι για το 2019-2020. Επίσης, ε, επικύρωσαν την ε, ενημερωμένη, ε, το ενημερωμένο σημείο της Τζούρι για τον αρχόν για περιπτώσεις ασυλίας και αποφάσισαν για μια μερομηνία για μια συζήτηση για τα θέματα σύγκρουση συμφερόντων την επόμενη εβδομάδα, 12 Νοεμβρίου. Και αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και περαιτέρω συζητήσει 14 και 14 Νοεμβρίου για το ίδιο θέμα μέσω γραπτή διαδικασία που ολοκληρώθηκε 9 Οκτωβρίου 2019, οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι τα εξή μέλη τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα είναι εκπρόσωποι τη Επιτροπή στι συναντήσει του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τι παραβιάσει θεματικών δικαιωμάτων. Κύριο Άξελ Βό, η κυρία ο κύριο Ιμπαν Καρθία Δελκάντο, ο κύριο Στεφάν Σεζουγνέ, ο κύριο Πάτρικ Μπρέγκ και ο κύριο Ζουλ Λεβοετό. γραπτή διαδικασία που ολοκληρώθηκε 10 Οκτωβρίου 2019, οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι για το πρώτο εξάμεινο του 2020 θα οργανωθεί μία ακρόαση για την ασφαλή, ιδεολογική και αποτελεσματική ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που θα έχει και χωριστά θέματα για τα θέματα ιδεολογίας και τα νομικά θέματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση ε, προσώπων, των, ε, δηλαδή των χαρακτηριστικών του προσώπου των ατόμων. Να κάνουν μία ε, αποστολή στο Λουξεμβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να έχουν μια συνεδρία στην Εθνικά Κοινοβούλια για να δοθεί το καλό παράδειγμα για καλύτερη νομοθέτηση από πλευρά ψηφιακή. Και επίση συμφώνησαν τι εκθέσει πρωτοβουλίε για τον τομέα τη ειδική πρωτοβουλία. Αποφάσισαν να προτείνουν στην ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών τι εξή προτάσει για προτάσει ίδια πρωτοβουλία. Δύο αιτήματα για νομοθετικέ εκθέσει ίδια πρωτοβουλία. Μία για τον ρυθμιστικό πλαίσιο για τι πλευρέ οντολογία τη τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τι σχετικέ τεχνολογίε και μία για το καθεστώς εθνικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη. Και δύο αιτήματα για συνήθεις ε, διαδικασίες ίδιες πρωτοβουλίες, για τα δικαιώματα πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα θέματα για της τεχνητή νοημοσύνης που σχετίζονται με την ερμηνεία, την ε, ε, εξουσία του κράτους και το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση. Συγγνώμη, ήταν πολλές οι ανακοινώσει. Το σημείο 4. Έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδρήσεων. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση, τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη 10η, 15η και 24η Ιουλίου 2019, 3η, 19η, 25-26 και 30 Σεπτεμβρίου 2019 και 14 Οκτωβρίου 2019, θα θεωρηθεί ότι ενεκρίθησαν. Έχει κανεί σχόλια από αυτών των πρακτικών. Σε αυτή τη φάση. Όχι. Λοιπόν, εάν έχετε σχόλια, μπορείτε να τα υποβάλλετε αργότερα. Θα εγκριθούν τα πρακτικά αυτά στο τέλο τη συνεδρία. Και τώρα, επειδή έχει αναβληθεί το 5, περνάμε στο σημείο 6, που είναι η παρουσίαση από τον Πασκάλ Λεαρντίνη, που είναι αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τον Βίλιαμ Σλίτ, που είναι διευθυντή στη Γενική Γραμματεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί των εξή θεμάτων. Ανακοίνωση τη Επιτροπή. Ανακοίνωση τη Επιτροπή, τη 15 η Τετάρτου 2019 για καλύτερη νομοθέτηση, Απολογισμό και επιμονή. Ανακοίνωση 23 Δεκάτου 2018, αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ενίσχυση του ρόλου των στην δημαμόρφωση τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση τη Επιτροπή 4 Εβδόμου 2019 για την επιτήρηση τη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ετήσια έκθεση και ανακοίνωση τη 17 Εβδόμου 2019 για την ενίσχυση του κράτου δικαίου εντό τη Ένωση ε, μια πρόταση δράση. Η Επιτροπή έχει καλέσει την Επιτροπή σε μια ανταλλαγή απόψεων για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα, την καλύτερη νομοθέτηση, την επιτήρηση τη εφαρμογή του νόμου τη Ένωση και το κράτο δικαίου. Η παρουσίαση από την Επιτροπή σήμερα θα βασιστεί στα πρόσφατα έγγραφα που ενέκρινε η Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Η συζήτηση θα είναι πολύ χρήσιμη για την περαιτέρω εργασία τη Επιτροπή μα για τα θέματα αυτά. Και ε, θέλω να ευχαριστήσω του δύο μιλητέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, δέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Από ό,τι κατάλαβα, η παρουσίαση του κυρίου Λεαρντίνη θα ασχοληθεί κυρίως με τα θέματα της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της καλύτερης νομοθέτησης, ενώ ο κύριος Σλίθ θα ασχοληθεί με το κράτος δικαίου και την εφαρμογή μεταξύ του κράτους δικαίου και της επιτήρησης της εφαρμογής του, του ενωσιακού νόμου από τα κράτη-μέλη. Θα έχετε 20 λεπτά. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε και μετά από τι παρουσιάσει αυτέ θα έχουμε ερωταπαντήσεις. Αυτό αναμένεται. Άρεστα ευχαριστώ πολύ. Οπότε, κύριε Ανεπροδοτή Γενική Διευθυντά, κύριε Λεαρντίνη, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε διαφορετικές επιτυχίες της ε, νομοθετικής διαδικασίας, νόμου παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ε, κάνοντα κάποιε αναφορέ στην επικουρικότητα, στην αναλογικότητα αλλά και στη βελτίωση τη νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά καταρχήν την επικουρικότητα, την αρχή τη επικουρικότητα, ε, σκοπεύει, στοχεύει μάλλον στο να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όσο το δυνατόν εγκύτερα στου πολίτε ε, και επίση στοχεύει στο να διασφαλίζει ότι η δράση που αναλαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη για να συμπληρώσει τα όσα συμβαίνουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ε, αυτή λοιπόν η αρχή, η οποία εφαρμόζεται στι μεικτέ αρμοδιότητε τη Ένωση με τα κράτη-μέλη, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλαμβάνει δράση ε, παρά μόνο στι περιπτώσει εκείνε όπου η ανάληψη κοινή δράση, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πιο αποτελεσματική από την ανάληψη δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Και ακριβώ επειδή έχει προστιθέμενη αξία η δραστηριοποίηση σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ε, αρχή λοιπόν, αρχή τη επικουρικότητα συνδέεται άρρηκτα και με την αρχή τη αναλογικότητα, η οποία σημαίνει ότι οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει του στόχου οι οποίοι έχουν θεσπιστεί στι συνθήκε εφαρμόζουμε εμείς από την πλευρά μας αυτές τις δύο αρχές και κατά την φάση της παραγωγής της νομοθεσίας αλλά και στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας. Δηλαδή όλες οι νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοδεύονται από μια αξιολόγηση αντικτύπου. Η αξιολόγηση αντικτύπου λοιπόν περιλαμβάνει και τα πορίσματα και τα όσα έχουν διαπιστωθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης η οποία προηγείται. Και στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης ε, τίθεται πάντοτε το ερώτημα του γιατί θα πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Πάντοτε λοιπόν ε, διασφαλίζουμε το ότι θα πρέπει να εξηγείται το γιατί χρειάζεται να αναλυφθεί δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και μετά, όταν έχει ήδη θεσπιστεί η νομοθεσία και βρισκόμαστε στη φάση της αναθεώρησής της, προβαίνουμε σε Διαδικασία αξιολόγηση στο πλαίσιο των οποίων πάντοτε ένα από τα πέντε βασικά κριτήρια είναι ακριβώ η προστιθέμενη αξία τη εν λόγω νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλι τώρα υιοθετηθεί από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρόταση δική τη, εξαρτάται από τα εθνικά κοινοβούλια η εξέταση του κατά πόσο τηρείται η αρχή τη επικουρικότητα με βάση και το πρωτόκολλο 2 στι συνθήκε. Έτσι λοιπόν, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δική τους άποψη και εφόσον το 1 τρίτο εκπροσωπεί τους, ε, υπάρχει εκπροσώπηση του 1 τρίτου από τις συνολικά 56 ψήφους, ε, τότε υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση της ε, αρχής της αναλογικότητας και εκεί υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει τη διαδικασία και έχει τη δυνατότητα είτε να επιμείνει σε αυτή την πρόταση αναδετυπώνοντάς την ή ε, αποσύροντάς την, αλλά πάντοτε θα πρέπει να δικαιολογήσει την απόφασή της αυτή. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω κάποιους αριθμούς εδώ, κάποια νούμερα ως προς το πώς ακριβώς λαμβάνει η χώρα αυτή η συνεργασία, αυτή η διαδίδαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε ό,τι αφορά καταρχήν τη γενική ανταλλαγή απόψεων ε, ανάμεσα στην Επιτροπή και τα Εθνικά Κοινοβούλια, να πούμε ότι ε, κατά τα τελευταία χρόνια ε, λαμβάνουμε 500 γνωμοδοτήσεις από Εθνικά Κοινοβούλια ετησίως. Ε, συνήθως λαμβάνουμε ε, λιγότερες ε, γνωμοδοτήσεις κατά την, το πρώτο έτος θητείας μιας επιτροπής κατά το τελευταίο έτος, ενώ μέσα στη μέση μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και στις 600 γνωμοδοτήσεις και βέβαια μπορούν να αφορούν όλα τα ζητήματα. Και τι σημαίνει αυτό, αν το διαιρέσουμε ανά τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, 20 περίπου γνωμοδοτήσει ανά κράτο μέλο. Από αυτέ λοιπόν τι 500 περίπου γνωμοδοτήσει που λαμβάνουμε ετησίω από το Εθνικά Κοινοβούλιο, κατά μέσο όρο υπάρχουν 30 από αυτέ οι οποίε αναφέρονται σε ζητήματα επικουρικότητα. Άρα λοιπόν αρκετέ, αλλά όχι επαρκή έτσι ώστε να οδηγήσουν ακριβώ στην ενεργοποίηση τη διαδικασία τη κίτρινη κάρτα ε, που ανέφερα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση δηλαδή νομοθεσία. Και κατά τα τελευταία πέντε έτη υπήρξε μόνο μία περίπτωση στο πλαίσιο τη οποία ακριβώ ενεργοποιήθηκε η διαδικασία τη ε, κίτρινη κάρτα. Πρόκειται δηλαδή για την αναθεώρηση τη οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Η μόνη λοιπόν κίτρινη κάρτα η οποία εφαρμόστηκε ω διαδικασία στο πλαίσιο τη Επιτροπή Juncker και εμεί επιμείναμε στη δική μα πρόταση δίνοντα εξηγήσει ε, και εξηγώντα αυτούς τους λόγους δηλαδή για την ε, επιμονή μας. Και στις 26 Ιουνίου του 2018 έγινε δεκτή τελικά από τους συνομοθέτες η αναθεωρημένη ε, πρόταση για την ε, αναδιατύπωση της οδηγίας. Άρα λοιπόν με αυτόν τον ε, τρόπο βλέπετε το πώ ενσωματώνεται η τήρηση αυτή της αρχής της ε, επικορικότητας στο πλαίσιο του διαλόγου της Επιτροπής με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα, το 2016, ο Πρόεδρος ε, Γιούνκερ δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για την τήρηση της αρχής της επικορικότητας τη αναλογικότητας και τη πιο αποτελεσματική ανάληψη δράση. Η ομάδα λοιπόν αυτή προέβησε κάποιες συστάσεις και τον Οκτώβριο του 2018 υιοθέτησε η Επιτροπή μία ανακοίνωση, την οποία αναφέρατε εσεί, κυρία Πρόεδρε, μόλι ε, τώρα, στην οποία εξηγούμε το πώ ακριβώ θα εφαρμόσουμε στην πράξη τι συστάσει αυτή τη ομάδα εργασία. Μία από αυτέ είναι ότι θα ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τι αρχέ τη επικουρικότητα και αναλογικότητα, με τυποποιημένο ε, τρόπο. Δηλαδή, μια τυποποιημένη διαδικασία αξιολόγηση, ειδικότερα τη ε, επικουρικότητα. Δηλαδή, θα εξετάζουμε συστηματικά τα ζητήματα που αφορούν την τήρηση αυτή τη αρχή σε όλε μα τι νομοθετικέ ε, και ελπίζουμε πως ε, το Συμβούλιο, το, το Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα χρησιμοποιήσουν αυτή την τυποποιημένη διαδικασία που δημιουργήσαμε για να διευκολύνουμε την εν λόγω διαδικασία. Επίσης, ε, στοχεύουμε ε, στην καλύτερη συμπερίληψη στη διαδικασία διαβούλευση των εθνικών και τοπικών και περιφερειακών αρχών, γιατί είναι και οι κύριοι χρήστε, αν θέλετε, αποδέκτε δηλαδή αυτή τη νομοθεσία και έχουν και άμεση εμπειρία τη εφαρμογή τη ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ένα τρίτο ε, σημείο είναι το ότι θα εξετάσουμε την ισχύουσα νομοθεσία έτσι ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και ποιος είναι ο ρόλος των περιφερειακών αρχών. Και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία Υπάρχει και το ζήτημα του πόσο μεγάλη χρονική προθεσμία δίνουμε στα εθνικά κοινοβούλια για να παρέμβουν, στο πλαίσιο δηλαδή τη διαδικασία του πρωτοκόλου 2. Οχτώ εβδομάδε ε, προβλέπονται, ε, αλλά εδώ έχουμε. πλέον συμπεριλαμβάνουμε υπόψη μας, δηλαδή σε αυτές τις 8 εβδομάδες λαμβάνουμε πλέον υπόψη μας ε, και την, ε, τις διαδικασίες που δεν λειτουργούν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Από εκεί και μετά θέλαμε να τονίσουμε και κάποιες από τις γνωδοτήσεις των ε, Εθνικών ε, Κοινοβουλίων και να τους δώσουμε δηλαδή ιδιαίτερη έμφαση ακόμα και αν ο αριθμός τους δεν ήταν επαρκής για να ενεργοποιήσει την κίτρινη κάρτα. Όπως σας εξήγησα μόλις τώρα, είναι σπάνια η περίπτωση όπου πράγματι φτάνουμε στο 1 τρίτο ε, των τοποθετήσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά αποφασίσαμε ότι εάν υπάρξει πράγματι κρίσιμη μάζα χωρίς να φτάνουμε στην κίτρινη κάρτα, δηλαδή τουλάχιστον 7 γνωμοδοτήσεις από 4 εθνικά κοινοβούλια, ε, θα δίδεται ιδιαίτερη ορατότητα, δηλαδή ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα με μια ε, απάντηση προς όλα αυτά τα εθνικά κοινοβούλια ε, σε λογική, εξεγώντας τους λόγους και δημοσιεύοντας την ελόγω τοποθέτησή μας ε, στο ευρύ απέναντι στο ευρύ κοινό και στου ε, συνομοθέτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την βελτίωση τη νομοθεσία, γνωρίζετε πω έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο στο πλαίσιο τη Επιτροπή Γιούνκερ και έχουμε δημιουργήσει τρεις ε, πυλώνες, διαβούλευση, αξιολόγηση αντικτύπου και αξιολόγηση ε, και αυτά τα στοιχεία θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας που θα εφαρμόζεται στο πλαίσιο δηλαδή της νομοθεσίας υπό την Επιτροπή Φοντερ Λάιεν. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει διαφανής νομοθετική ε, διαδικασία στην οποία θα περιλαμβάνονται οι πολίτες και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς. Και στο πρόσφατο Regulatory Policy Outlook του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήθηκε πως στο πλαίσιο των ε, μοχωνών που ε, συμμετέχουν ε, στον ΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέχει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά αυτή την αξιολόγηση τη νομοθεσία. Επίση, είμαστε ανέκαθεν υπέρ του one in, one out, αυτή την αρχή δηλαδή τη υιοθέτηση νέα νομοθεσία στο βαθμό που Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κίνητρα έτσι ώστε να εξετάζουμε πάντοτε την ισχύουσα νομοθεσία και να διαπιστώνουμε πού υπάρχουν περιθώρια να περικοπεί νομοθεσία όταν υιοθετείται καινούργια νομοθεσία. Και αυτός ο στόχος βέβαια εδώ είναι να μην ή να αντισταθμίζουμε τα, τα εμπόδια που ενδεχομένως να δημιουργεί η νέα νομοθεσία μέσω κατάργησης ε, άλλων εμποδίων τα οποία δημιουργούσε παλαιότερη νομοθεσία. Και ε, θα είμαστε και πιο συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής τη αρχή στο πλαίσιο του ε, προγράμματος εργασιών της ε, Επιτροπής για το 2020, το οποίο πρόγραμμα εργασιών θα υιοθετηθεί ε, λίγε εβδομάδε μετά από την επίσημη ανάλυση των καθηκόντων της Νέας Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας πούμε δύο λόγια όσον αφορά τις πρόσφατες εκθέσει για την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Πρόκειται για την αποτελεσματική εφαρμογή του που είναι πάρα πολύ ή ίσως και από τα πιο σημαντικά όσον αφορά την πολιτική της Ένωσης, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα που να μπορούν να σκεφτούν τα δικαιώματα, να μπορεί κανείς επίσης να την χάνει δικαστικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης αυτών και όπως είπε ο προλαλής σας, πρόεδρος, Πάρα πολλά από αυτά τα θέματα έχουν επικάλυψη με την υπόθεση του κράτους δικαίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επομένω ότι εφαρμόζεται ο νόμος, ότι υπάρχει συμμόρφωση, είναι υψηλή προτεραιότητα και για την επιτροπή αυτή, αλλά και στις κατευθυντήριες γραμμές γιατί αυτό της νεοεκλεγήσης, τη Πρόεδρο και ε, ακόμη για να έχουμε αυτή την ετήσια έκθεση όσον αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία τη εφαρμογή του κοινωνικού δικαίου, έχουμε μια γενική έποψη για το τι έγινε το 2018. Επίση όμω όλα αυτά ε, αντικατοπτρίζουν μια μακρόπνοη, μακροπρόθεσμη τάση και ελπίζουμε ότι ε, θα συνεχιστεί αυτή η τάση και στο μέλλον. Τρία να θα ήθελα να θίξω. Πρώτα-πρώτα αυτή η έκθεση αναδεικνύεται ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της δράσης για, για, την εξασφάλιση δηλαδή της εφαρμογής του κοινωνικού δικαίου και των προτεραιών για τις πολιτικές μας και οι βασικές πολιτικές εκεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής του κοινωνικού δικαίου είναι οι εξή πολιτικές περιβάλλον, πολιτικές αυτά δηλαδή που καίνε τους πολίτες αλλά και τα θέματα της ιστορικής αγοράς αλλά σε κάθε τομέα προτεραιότητα βλέπουμε το ότι οι συγκεκριμένε δράσει έχουν πραγματικέ επιπτώσει όσον αφορά την υλοποίηση τη κάθε πολιτική. Βλέπουμε δηλαδή πόσο άμεση σχέση έχει η ορθή εφαρμογή του δικαίου και η επιπτώσει αυτού. Επίση, βλέποντα στην έκθεση ότι δεν αναφέρονται μόνο οι παραβάσει, αλλά και το θέμα της πρόληψης, διότι από το 2014 είχαμε 90% των ε, ε, υποθέσεων παραβίασης του δικαίου που εξετάστηκαν χωρίς να υπάρχει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και έτσι είχαμε εξοικονόμηση χρημάτων των φορολογουμένων και αυτό είναι απότοκο του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ τη Επιτροπή και των κρατών ε, μελών. Οπότε έχουμε ένα σωρό τώρα μέσα και εργαλεία, ούτω ώστε μπορούμε να βοηθήσουμε τα κρατημέλη να μεταφέρουν στο ιστορικό δίκαιο, να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν τα όσα προβλέπει το κοινωτικό δίκαιο ορθώς και εγκαίρως εργαστήρια, κατάρτιση και κατευθυντήριες. Τέλος, αυτή η έκθεση λεπτομερώς εξηγεί, όπως και σε άλλες εκθέσεις, εξηγείται τι κάνουμε στις ε, περιπτώσεις των παραβάσεων του δικαίου και καταγγελιώνω το ώστε να δώσουμε μια συνέχεια στα όσα επισημαίνει ο διαμεσολαβητής αλλά και το ελληνικό συνέδριο. Εδώ δίνει και το θέμα βέβαια το πόσο χρόνο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ερευνήσει τις πιθανές παραβάσεις. Συνολικά, είχαμε κορύφωση των στοιχείων το 2016 και μετά το 2018 είχαμε μια μικρή πτώση κατά 5% σε σχέση με το 2016. Έχουμε και άλλα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη μετέφεραν τις ε, οδηγίες το 2018 συντομότερα από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά ο αριθμός των καταγγελιών ακόμη είναι υψηλός και τελικά αυτό που έγινε την έκθεση είναι το ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπαθίες μας τόσο ώστε να ενημερώνουμε τους πολίτες για τα δικαιώματα και για τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Έτσι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί το κράτος δικαίου και πάμε τώρα. Σε πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου. Κάποιες διαδικασίες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Βέβαια αυτό είναι ο πυρήνας των αξιών μας. Είναι στο επίκεντρο αυτό, όπως το άρθρο 2 της συνθήκης προβλέπει. Και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή του δικαίου και ε, εδώ είναι το θεμέλιο της αμοιβαία εμπιστοσύνη που ακριβώς ε, είναι το θεμέλιο του ευρωπαϊκού οραματο, Οπότε θα να δούμε το ότι εδώ έχουμε τις προτεραιότητες, ε, από εδώ δηλαδή πηγάζουν για τα τρία θεσμικά όργανα και το ευρωβαράμετρο φέτο φέτος κατέληξε στο ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ κόσμος για όλα αυτά. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόσφατα κατέληξε στο ότι το κρατός δικαίου και πιο συγκεκριμένα η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό βαθμία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει αυτή την εργαλειοθήκη όπως λέμε για να υλοποιήσει το κράτος δικαίου και αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια και έχουμε τι προτάσει τη ε, ανακοίνωσή μα του Ιουλίου. Αλλά επίση έχουμε και τι ε, κατευθυντήριες τη ε, Προέδρου που είναι ακόμη ένα βήμα ούτω ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η εργαλειοθήκη και συγκεκριμένα τώρα έχουμε μια ευρύτερη βεντάλια από δράση ώστε να καλύψουμε και να διαδώσουμε αυτό, αυτό το πνεύμα του κράτους δικαίου, να προλάβουμε τα προβλήματα και εκ των υστέρων όταν προκύψουν να τα λύσουμε. Οπότε αυτού του είδους το πνεύμα, αυτή η κουλτούρα ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει προβληματική, διάλογος, κοινωνία των πολιτών, και, αλλά και να εμπλακούν σε αυτό και φορείς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οπότε και η Επιτροπή σας σε αυτά τα πλαίσια είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει. Αυτός ο κύκλος των προσπαθειών για το κράτος δικαίου κορυφώθηκε σε αυτή την ε, έκθεση που θέλουμε να δούμε εδώ τι μπορεί να γίνει ως εργαλείο πρόληψης και θέλουμε να υπάρχει κάποιο είδους ε, ανταλλαγή στοιχείων, να υπάρχει διάλογος από όλες τις πλευρές και αυτό ακριβώς θα αναδείξει καλύτερε πρακτικέ και θα επισημάνει τα βασικότερα προβλήματα. Αλλά η Επιτροπή, όπω και το Συμβούλιο, ελπίζει ότι με την έκθεση αυτή θα βοηθήσουμε και το δικό σα έργο του Κοινοβουλίου σε αυτή την ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος είναι το ότι θα πρέπει να παρεμβαίνει ε, λιγότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να προσφύγει στα διάφορα που περιέχει αυτή η εργαλειοθήκη του κράτου δικαίου ούτω ώστε να υπάρχει αποκλιμάκωση και επίσης η κατάσταση να αποκαθίσταται σε μια κανονικότητα. Και όλα αυτά επί τη βάση κάποιων βασικών αρχών, για παράδειγμα, τα κρατημέλη θα πρέπει εξίσου να εμπλέκονται η βασική ευθύνη και αρμοδιότητα είναι το κρατών μελών και ότι κανείς θα πρέπει πρώτα απ' να χρησιμοποιεί την ε, προσέγγιση του κράτους δικαίου και τους μηχανισμούς ε, του εθνικού δικαίου. Οπότε έτσι θα πρέπει να κάνουμε βήματα πρόοδο με συνεργασία. Τέλος, είναι κοινή προσπάθεια τα εν λόγω όλα τα θεσμικά για τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν αυτέ τι εγγύσει για την τήρηση του κράτου δικαίου. Και είναι πιο αποτελεσματική από το για αυτή τη προσπάθεια όταν υπάρχει συνοσμό μεταξύ των ε, διαφόρων θεσμικών οργάνων. Και γι' αυτό αυτή η έκθεση του εξαδρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, οργάνωση στο ότι θα γίνει, ούτω ώστε να εμπλέκονται όλα τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος θαυμάσεις και σαφέστατε ε, παρουσιάσεις, όπως συνήθω. Υπάρχουν ερωτήσεις ε, από τους συναδέλφους. Ναι, για κύριε τους δύο, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ για τις εκθέσεις σας, τις παρουσιάσεις σας. Τώρα εγώ ενδιαφέρομαι για την καλύτερη νομοθέτηση. Θαυμάσια συνόψη. Και επίσης μας παρουσιάσετε και τις νέες συστάσεις. Να ρωτήσω το εξής. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι πολύ σημαντικό. Καθώς και τα διάφορα επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις να συμμετέχουν περισσότερο στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Και η Επιτροπή Περιφερειών θα μπορούσε να παίξει ρόλο σε αυτό λοιπόν. Οι γνωμοδοτήσεις τη βέβαια δεν είναι δεσμευτικέ αλλά λαμβάνονται υπόψη. Έχετε συζητήσεις στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι προτάσεις της Επιτροπής Περιφερειών το οποίο όπως ξέρετε αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από δημάρχους, ε, συμβούλους, ε, δημοτικούς, ε, κοινοτικούς, περιφερειακούς. Αυτό θα αύξανε την αποτελεσματικότητα και της νομοθέτησης και της εφαρμογής. Από τη διαδικασία λοιπόν διαβούλευσης της, που είχατε με την Επιτροπή Περιφερειών προέκυψε κάτι το θετικό για την νομοθέτησή σας και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει απλώς έτσι, τυπικές σχέσεις με την Επιτροπή Περιφερειών. Ξέρετε, οι συνθήκες λένε ότι πρέπει να γνωμοδοτεί για τις νομοθετικές προτάσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτεί και το δεύτερο η Επιτροπή Περιφερειών έχει πολύ ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να προσφύγει κατά της Επιτροπής στη δικαιοσύνη για παράβαση της αρχής επικουρικότητας. Είναι βέβαια ε, η λύση χρήσης πυρηνικών όπλων αυτή που δεν έχει χρειαστεί να αξιοποιηθεί μέχρι τώρα λόγω του διαλόγου. Επίσης ε, η Επιτροπή Περιφερειών και πολλά συγκεκριμένα μέλη από διάφορες περιφέρειες και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστούν το παρατηρητήριο για την επικουρικότητα και μπορούν να μας ε, ειδοποιήσουν εγκαίρως αν υπάρχουν προβλήματα επ' αυτού. Και κατά τη διετία της αυτή η Επιτροπή έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα REFIT, αναδιατύπωση. Εκεί υπάρχουν εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη και από άλλους ε, φορείς, ε, επιχειρήσεις, συνδικάτα, κοινωνία των πολιτών, και άλλους για να εντοπίσουμε νομοθετήματα που δεν εφαρμόζονται σωστά και η Επιτροπή Περιφερειών έχει, είναι πλήρες, πλήρες μέλος σε αυτό το παρατηρητήριο. Μπορούν να ε, ενημερώσουν την πλατφόρμα Refit αν υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη γνώμη τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Λεπρετών σε και μετά εσείς, παρακαλώ. Κύριε Λεπρετών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάφορες παρατηρήσεις έχω να κάνω. Τα κείμενα είναι μακροσκελή και οι παρουσίες που μας έγινε επίσης. Παρουσιάσεις. Τώρα για την επικουρικότητα. Άκουσα με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Κατά μέσο όρο κάθε χρόνο κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο στέλνει 30 αναφορές για επικουρικότητα. Εντάξει δεν είναι τρομερό αλλά αξιοσημείωτο και τα πέντε τελευταία χρόνια μόνο μια κίτρινη κάρτα βγήκε. Και το θυμόμαστε όλοι γιατί ήταν ένα θέμα που είχε μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη, αναθεώρηση οδηγία για του ε, αποσπασμένου εργαζόμενου. Αλλά δεν έγινε τίποτα διότι η Επιτροπή τελικά ε, ε, επέμενε στη θέση τη. Τι κάνετε για να βελτιωθεί ο σεβασμός της επικουρικότητας. Με ενδιαφέρει πολύ. Ναι, αυτά που είπατε αποδεικνύουν ότι κάτι κάνετε. Αλλά πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτός ο πίνακας για την ε, αξιολόγηση της επικουρικότητας. Καλή προσπάθεια. Είναι ένα εργαλείο εύχριστο που επιτρέπει σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια να επιχειρήσουν να έχουν τα ίδια κριτήρια για να κρίνουν πώ εφαρμόζεται η επικουρικότητα. Και το άλλο που είναι και πιο ενδιαφέρον είναι αυτή η βούληση να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι γνώμες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και όπως είπατε και εσείς τώρα, δυστυχώ δεν τα πάει πολύ καλά η κίτρινη κάρτα. Οπότε, αυτό που λέτε ότι όταν τέσσερα Εθνικά Κοινοβούλια επικρίνουν ένα νομοθέτημα, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να απαντήσει αιτιολογημένα στις ανησυχίες τους. Είναι ας πούμε μια μίνι κίτρινη κάρτα. Ενδιαφέρον είναι αρκετά ευέλικτο όργανο. Κάτι άλλο που δεν το είπατε, αλλά είναι στα έγγραφα. Είπατε ότι θα επιμηκύνετε τις προθεσμίες για να προσπαθήσουν να απαντήσουν, να αντιδράσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα είναι 8 εβδομάδες, θέλετε να γίνει 12. Ναι, συμφωνώ. Θα επέτρεπε να λυθούν τα προβλήματα, ξέρω εγώ, καλοκαίρι, Χριστούγεννα κτλ. Τέλος αφού σας επένεσα, τώρα θα σας επικρίνω κιόλα, κιόλας, αλλά μην ανησυχείτε. Έχω ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα, η επικουρικότητα δεν εφαρμόζεται πολύ καλά και είναι αναπόφευκτο. Γιατί είναι και δικαστής και διάδικος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι κάναμε λάθος. Θυμάμαι τις συζητήσεις που κάναμε στη Γαλλία όταν εγκρίναμε την συνθήκη του Μαστρίχτ που εισήγαγε στο 3β άρθρο την επικουρικότητα. Και λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να μπορεί να αποδείξει κάθε φορά ότι ε, μπορεί να δράσει καλύτερα από τα κράτη-μέλη για κάποιο θέμα. Αλλά στην ουσία ισχύει το αντίστροφο. Αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πού θα δράσει και κατόπιν τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να αποδείξουν ότι εκείνα θα ήταν πιο κατάλληλο να ασχοληθούν με το ΑΒ θέμα. Νομίζω ότι έχει αντιστραφεί λοιπόν η αρχή της επικουρικότητας. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση, το αντιλαμβάνεστε ότι έτσι το αισθάνονται οι πολίτες, ότι έχει αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης. Και κάτι που με ενδιαφέρει πολύ ε, πιο συγκεκριμένα, ίσως γιατί μεγάλος, ε, αναμφίβολα γιατί μεγάλος, ε, είναι ένα πολύ συγκεντρωτικό κράτος για μένα, η επικουρικότητα είναι όπλο κατά της εθνικής κυριαρχίας. Αξιοποιείται η, κυριαρχία, η επικουρικότητα για να υπάρχει απευθείας διάλογος μεταξύ των περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βραχικυκλώνοντας τα κράτη. Και αν ε, αμφιβάλλετε, διαβάστε ε, στη σελίδα 14, την τελευταία σελίδα του κειμένου που μας δόθηκε. Εκεί, σε αυτό το πίνακα με γκρι φόντο, υπάρχει αυτή η φράση. Η Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει να δημιουργήσει περιφερειακού πόλου που να επιτρέπουν να γίνεται πιο αποτελεσματική μεταφορά της πείρας των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε αυτού που αποφασίζουν για ε, την πολιτική τη Ένωση. Εδώ απλώ εξαιρούμε τα κράτη-μέλη. Για μένα δεν είναι σωστό αυτό. Αυτή λοιπόν η δεύτερη ερώτηση λοιπόν, που θέλω να θέσω. Αναγνωρίζετε ότι η επικουρικότητα μπορεί τελικά να αξιοποιηθεί για να εξαιρεθεί από την συζήτηση το κράτο μέλο. Τώρα για το δεύτερο έγγραφο, για την ενίσχυση του κράτου δικαίου, μια πολύ σύντομη ενημέρωση, κάτι που, για το οποίο θέλω να σε ενημερώσω. Το έγγραφο για τον έλεγχο τη εφαρμογή του δικαίου. Στη σελίδα 5 λέγεται ότι η Γαλλία διώκεται γιατί δεν ε, σέβεται την νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα. Εδώ και λίγες μέρες καταδικάστηκε, όχι απλώς ε, διώκεται. Ε, στο Παρίσι συμφωνήθηκε η συμφωνία για το κλίμα και καταδικαζόμαστε για την ποιότητα του αέρα και για το κράτος δικαίου. Στο έγγραφο που μας εστάλει και που είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπενθυμίζει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κράτου δικαίου. Εγώ θα τα είχα παρουσιάσει αλλιώ. Θα έλεγα ότι το κράτο δικαίου είναι ε, τυπικό θέμα, είναι η ιεράρχηση των νόμων, ενώ το ουσιώδε θέμα είναι ο σεβασμό των αξιών. Και μεταξύ των αξιών αυτών αναφέρεται ο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Χαίρομαι γιατί αυτό υπερασπιζόμαστε, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Και μια επίκριση. Εκπλήσουμε πάντα όταν ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι, λέει ότι είναι κράτος δικαίου. <clears throat> Μα πώς μπορεί να είναι κράτος δικαίου αφού δεν είναι κράτος. Είναι λάθος χρήση όρονα. Οπότε ερώτηση. <clears throat> Το αναγνωρίζετε ότι δεν είναι σωστή η χρήση αυτού του όρου. <clears throat> Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλον. Σκέφτεστε ποιον. Και κάτι ακόμη. Δεν έχετε την εντύπωση ότι αυτή η έννοια του κράτους δικαίου τελικά αξιοποιείται για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η υπεροχή της Ένωσης επί των κρατών μελών. Και αυτό επιβεβαιώνεται στην τελευταία σελίδα, όπου συνήθως λέμε τα πράγματα στα ράτα, στην τελευταία σελίδα λέμε ότι για να γίνει καλύτερα σεβαστό το κράτος δικαίου προτείνεται να δημιουργήσετε και νέους μηχανισμούς κυρώσεων για τα κράτη-μέλη που θα θεωρηθεί ότι δεν σέβονται επαρκώς το κράτος δικαίου. Εδώ δεν πρόκειται για το άρθρο 7 του, της συνθήκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται να επινοήσετε και άλλους μηχανισμούς. Αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Βεβαίως με ενδιαφέρει το κράτος δικαίου. Αλλά για να γίνεται σεβαστό πρέπει να ε, επιλέγουμε την συνεργασία, όχι τις κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ δείξατε μία φορά μία σειρά από ζητήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω τώρα να αρχίσουμε φιλοσοφική συζήτηση για το κατά πόσον η αρχή της επικουρικότητας είναι πολιτική έννοια ή κοινωνιολογική, γιατί τώρα μιλούμε ε, νομικά και έχουμε ακριβώς όλο το νομικό πλέγμα που διαπνέει τη συνθήκη που ορίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων, της Επιτροπής των Περιφερειών, τέλος πάντων ο καθένας τις δικές του αρμοδιότητες. Οπότε βέβαια υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την τήρηση της αρχής υπηγουρικότητας και ε, για την ενδεχόμενη χρήση της κεντρικής κάρτας, για τις περιφέρειες, για δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο. Είναι μια σειρά διατάξεων που έχουν χαρακτήρα νομικό. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια εκείνο βέβαια πολλές φορές ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια διατυπώνουν κάποιες απόψεις όσον αφορά ε, το, το, το, πλαίσιο του σεβασμού. Ε, και όμως δεν είναι το θέμα του πλαισίου, είναι θέμα της ουσίας. Δεν είναι το αν ε, μπορεί όχι να επέμβει η Κομισιόν, αλλά είναι το, το τι κατεύθυνση έχουν οι προτάσεις της Κομισιόν, τι χαρακτήρα έχουν. Άρα δεν έχουμε προκειμένου σεβασμό τήρηση της αρχής επικουρικότητας. Οπότε ας μείνουμε σε αυτά τα πλαίσια, τα νομοπαρασκευαστικά και στα όσα νομοθετικά προβλέπονται. Οπότε, εντάξει, είναι θέμα ε, ενημέρωσης, κατάρτισης. Δεν, δεν υπάρχει θέμα κατά κανενός. Άρα έτσι μπορεί να έχουμε αυτή την βοήθεια που αναφέρθηκε για την εφαρμογή στην καθημερινή ζωή του κοινοτικού δικαίου για τις, ε, το, τους διαγωνισμούς, ε, τις δημοπρασίες, τέλο πάντων. Αυτό τα ξέρουν οι τοπικές περιφερειακές αρχές. Ε, αυτοί ξέρουν τι ισχύει και τι προβλήματα υπάρχουν. Τώρα όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, εδώ υπάρχουν νομικά προβλήματα, ότι προβλέπεται 8 εβδομάδες και όχι παραπάνω η συνθήκη. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να χορηγηθούν 12 ε, εβδομάδες χωρίς να τροποποιήσουν το πρωτοκόλλο 2 αλλά μπορούν να όργανα να αφαιρέσουν από αυτό το δικαίωμα τις διακοπές χριστουγεννιάτικες, ε, ε, φερινές, ούτως ώστε να μείνουμε στο πλαίσιο των 8 καθαρών ημερών εργασίας, εβδομάδων εργασίας, των κοινοβουλίων. Σλίτ. Ακριβώς για το θέμα του κράτους του δικαίου. Ναι, ναι. Τα λέει η συνθήκη. Έχει ουσία αυτή η αρχή. Και είναι σημαντικό να το χωνέψουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε θα πρέπει να διοδοθεί αυτό το πνεύμα τήρησης του κράτους δικαίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μία κοινή αντιμετώπιση, κοινή κατανόηση. Τα είδαμε στις πρόσφατες ε, αποφάσεις, την πρόσφατη νομολογία, το τι σημασία έχει αυτή η κατανόηση από όλους. Πάντως θα πρέπει ακόμα να καταφέρουν προσπάθειες ούτως ώστε να είναι γενικότερη ευρύτερη αυτή η κατανόηση του περί τίνος πρόκειται. Επίσης, για την προσέγγιση. Γι' αυτό και επιμένει στις κατευθυντήριες της Προέδρου μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό τονίζουμε. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και διάλογος. Συνεργασία. Πρέπει ο κ. Λεμπρετό. Το ρίζει στο 7-4 η συνθήκη. Λέει πώ μπορούμε να ενεργούμε όταν προκύπτουν προβλήματα σε αυτή τη διάταξη που μας ανέφερε ορίζονται διάφορα που αφορούν συγκεκριμένες πολιτικές ένωσες και βέβαια χρειάζονται συμπληρωματικά και άλλα μέσα. Οπότε γι' αυτό και η Κομισιόν πως αυτή την πρόταση στα πλαίσια του, της δέσμες μέτρων για το πολιετές δημοσιομικό πλαίσιο και έτσι τα θέματα του κράτους δικαίου να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ίσως βέβαια και σε άλλους τομείς με στοχευμένο τρόπο. Εξετάσουμε να δούμε τι άλλα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα αυτά βέβαια θα περάσουν μέσα από την νομοθετική διαδικασία. Με αυτό το πνεύμα μέρος να ενεργούμε. Τη συνεργασία και κατανόηση αυτού του πνεύματος, αυτής της κουλτούρας του κράτους δικαίου. Και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για αυτές τις ε, διεξοδικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχουμε ε, τρεις ακόμα ομιλητέ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να του παρακαλέσω να είναι σύντομοι. Ο Σάγια καταρχήν. Σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ε, ε, ε το γεγονό ότι συζητούμε από κοινού αυτά τα τρία-τέσσερα ζητήματα, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αναφορά μέσα σε αυτά τα έγγραφα από το ένα ζήτημα στο άλλο. Ίσως ε, θα μπορούσε να υπάρχει με την ανακοίνωση. Δηλαδή, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Γίνεται μια αναφορά στη βελτίωση τη νομοθεσία και στην αξιολόγηση αντικτύπου για το γεγονό ότι ο στόχο αυτή τη αξιολόγηση αντικτύπου είναι η εξέταση του κατά πόσο η προτινόμενη πράξη εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, στο ίδιο ε, ζήτημα σε αυτό που νομοθετεί. Και μετά σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τη ε, σχετική ανακοίνωση γίνεται μια διαφορετική απάντηση. Δηλαδή γίνονται αναφορές σε ζητήματα οποία δεν αφορούν αμυγός ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πράγμα το οποίο δηλαδή ε, συνηγορεί προς το ότι όταν συζητούμε αυτά τα ζητήματα και ειδικότερα το ζήτημα του κράτους δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα παντού. Και τίθεται το ερώτημα του πώς ε, θα, θα, θα παράσουμε τις απαραίτητες εγγυήσεις προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, ειδικότερα αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, θεωρείται πως εκείνη θα πρέπει να διασφαλίζει ακριβώς την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Πώ όμω θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να εγγυηθούμε ότι εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα παντού με τον ίδιο τρόπο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, από τη δική μου χώρα ε, γίνονται πολλέ συζητήσει και εδώ και αλλού σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία ε, τη ε, δικαστική εξουσία. Ειδικότερα στη δική μου χώρα. Και από την άλλη πλευρά, όταν κάνει, κάνεις, ε, ρίχνει μια ματιά στο scoreboard, σε αυτό το πίνακα βαθμολογία σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτήν την δικαστική εξουσία, δεν απηχείται αυτή η ανησυχία εκεί. Δηλαδή, ε, είτε βρισκόμαστε κάπου στο μέσο όρο ή σε κάποια άλλα ζητήματα βρισκόμαστε ε, σε πολύ ψηλή βαθμολογία. Δηλαδή υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα της ε, ανεξαρτησίας του δικαστικού σωματού, τη Δικαστική εξουσία. Πώ λοιπόν, ερωτώ, μπορούμε να έχουμε την εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο προτύπων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση. γιατί αν δεν εφαρμόσουμε τα ίδια πρότυπα, ουσιαστικά επιλέγουμε εμείς αυτά που θέλουμε να κρίνουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την επικορικότητα και την αναλογικότητα, εδώ αποτελεί ε, πρόβλημα το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, ισορροπήσουμε καλύτερα, να εξετάσουμε λίγο καλύτερα το ζήτημα του κράτους δικαίου σε σχέση με αυτά τα δύο πρότυπα. Γιατί η συνθήκη αναφέρει ξεκάθαρα ότι το κράτος δικαίου δεν αφορά μόνο στα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη όλα τους διαθέτουν μηχανισμό λιγότερο ή περισσότερο ε, για την διασφάλιση αυτού του κράτους δικαίου, δηλαδή μέσω συνταγματικών δικαστηρίων και άλλων τέτοιων διαδικασιών που ε, διασφαλίζουν ακριβώς την τρίση του κράτους ε, δικαίου. Σε ελάχιστες περιπτώσεις δηλαδή χρειάζεται να υπερβούμε το εθνικό επίπεδο. Αντιθέτως όμως, όταν αναφερόμαστε στα θεσμικά όργανα της ίδιας της Ένωσης, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και ούτω καθεξής, και ελέγχουμε για παράδειγμα τα ζητήματα σύγκρουση συμφερόντων των επιτρόπων, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες ως προς το κατά πόσο εφαρμάζονται αυτά τα πρότυπα εδώ. Οπότε, όταν αναφερόμαστε στο μηχανισμό της διασφάλισης του κράτους δικαίου, θα πρέπει κάπου να αναφέρουμε ότι αυτή η αρχή του κράτους δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρότητα, αυστηρότερα και πολύ συγκεκριμένα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι δεν μπορεί δηλαδή να είναι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο ειδικότερα που έχει πολιτικό χαρακτήρα, που θα ε, κρίνει τα κράτη-μέλη. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει εδώ ένα πιο ήπιο μηχανισμό ε, ό,τι αφορά αυτή την αξιολόγηση των ε, κρατών σε σχέση με την τήρηση του κράτου δικαίου. Ε, θέτω λοιπόν το ερώτημα του πώ θα εφαρμόσουμε αυτέ τι αρχέ τη επικουρικότητα, τη αναλογικότητα και των ίδιων προτύπων για όλα τα κράτη-μέλη. Ειδικότερα όταν για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την εσωτερική συνταγματική τάξη ή τις νομοθετικές διαδικασίες των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Παρακαλώ οι μελητές μας ε, να δώσουν κάποιες απαντήσεις αν θέλουν σύντομα και μετά θα ακούσουμε τους δύο τελευταίους ομιλητές μας που έχουμε από τα μέλη. Ναι. Όταν κάνουμε λόγο για αναλογικότητα και επικορικότητα, κάνουμε πάντοτε λόγο για νέα νομοθεσία η οποία θα εφαρμόζεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν ε, το ζήτημα της εναρμόνισης σε ε, μικρότερο βαθμό αποτελεί πάντοτε ζήτημα που εξετάζει αξιολόγηση αντικτύπου γιατί πάντοτε θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και σωστά η νέα νομοθεσία. Ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει τόσο οξύ αν θέλετε χαρακτήρα αυτή την περίοδο είναι η φύση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ε, δηλαδή παλαιότερα αναφερόμασταν σε οδηγίες, σε πλαίσια ή πλήρους αναρμόνισης, ε, από εκεί και μετά σε κανονισμούς ε, και σε, κά... σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε νομικές πράξεις οι οποίες επιτρέπουν ακριβώ κάποια περιθώρια ευελιξία στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, τη μεταφορά αυτή τη νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε σε σχέση με την εθνική νομοθεσία σχέση δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά το κράτος ε, ε, ε, δικαίου, εξετάζουμε το πού βρίσκεται η εθνική νομοθεσία σε σχέση ακριβώς με την εφαρμογή του κράτους δικαίου ως έχει. Και εγώ να προσθέσω και να επαναλάβω αυτό που είπαμε ότι δηλαδή Η φιλοσοφία μας είναι ακριβώς η επικοινωνία και η αναγνώριση ότι το κάθε κράτος μέλος πράγματι διαθέτει τη δική του συνταγματική τάξη. Ε, οι οποίες διαφορετικές τάξεις ποτέ δεν είναι ίδιες μεταξύ τους, ε, δεν μπορούν να είναι πλήρως εναρμονισμένες και στο πλαίσιο των οποίων ε, υπάρχουν διαφορετικές εθνικές παραδόσεις. Όμως ισχύει ταυτόχρονα ότι αν θέλουμε να είμαστε, αν θέλουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και σημαίνει το ίδιο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, ε, τότε ναι, θα πρέπει να εξετάζουμε ακριβώς και αυτή την πτυχή του, της ύπαρξης του κράτους δικαίου στην Ένωση. Και... Για... Ακριβώς επανέρχομαι σε αυτό που αναφέρομαι ότι θα πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα με έναν τοπία κράτους δικαίου στην Ένωση. Που βέβαια δεν αποτελεί ένα ενίο πρότυπο. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για ένα τομέα στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες, αλλά πάντοτε ε, με συλλογικό τρόπο, συνεργαζόμενοι μεταξύ μας. Ευχαριστώ, λέει ε, Πρόεδρος. Ε, θα ακούσουμε και τους δύο τελευταίους ομιλητές μας ε, και στην συνέχεια θα απαντήσουν και πάλι παραλύσεις. Ο κ. Ε, είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε επίσης και για τα όσα μας εξηγήσατε. Να σας πω για την επικουρικότητα. Συμφωνώ με αυτό που μας είπατε. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής κουλτούρας στην ε, Ιταλία. Κάτι το οποίο προκύπτει διαχρονικά. Πέραν όλων των άλλων που σαφώς και συμφωνώ, έχω επισμένα ένα πρόβλημα. Θεωρείτε ότι αυτή η αρχή ακριβώς όπως διατυπώνεται και εγώ συμφωνώ, η αρχή της επικουρικότητας που Θέλω να πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μόνο αυτά τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε επίπεδο κυριαρχού αρχών, κρατών ή τοπικών αρχών. Θεωρείτε ότι έτσι πιάνει τόπο αυτή η αρχή. Το θέμα δεν είναι μια παραχωρήση πολιτικού επιπέδου είναι το ποιες είναι οι επιπτώσεις με το που εφαρμόζεται λίγο ή πολύ αυτή η αρχή. Της επικουρικότητας δεν προκύπτει αδιαστατότητα ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί, ίσως κακός, κάποιο είδους απέχθεια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φαίνεται ότι η Ευρώπη επιβάλλει κανόνες. Κανόνες που θα μπορούσαν να αφαιθούν στα κυρίαρχα κράτη ή στις τοπικές αρχές του κάθε κράτους μέλους. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αυτό το είδους η αντίφαση μεταξύ της θεωρίας και της ε, εφαρμογής της αρχής. Της μίας και της άλλης. Και αναλογικότητας και επικορικότητας. Αυτό λοιπόν φέρνει την αντίθεση από τον κόσμο. Οπότε και εμείς ως πολιτική αυτό θα πρέπει να θέσουμε. Ε, φυσικά και εμείς ε, είμαστε φιλευρωπαίοι, αλλά θα πρέπει αυτό να θέσουμε το πώς, πώς, μέσα και με τους κανόνες και μέσω της συγκεκριμένη υλοποίηση και εφαρμογή αρχής τη υποκριτικότητα, πώς θα μπορέσουμε να ανασχέσουμε, να φρενάρουμε αυτή την κοινή πεποίθηση, ότι συχνά, συχνά, αντίθετα με τους ίδιους τις τους στόχους Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς να το πω. Κάνει αντίθετα, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίο. Σε επίπεδο ηγεσία. Και προκύπτει αυτή η αντίθεση λοιπόν. Και αυτή υπάρχει αυτή η λεπτή διαφορά μεταξύ πολιτικής αρχής και εκτελεστικής. Άρα κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε αυτού του είδους το αρνητικό φαινόμενο να φρεναριστεί. Um, and, um, Jackie Jones. Finally in the right room and the right time. Ε, Jackie Jones έχει το λόγο. Επιτέλους βρίσκομαι σωστή, σωστή, σωστή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, αστείευομαι. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω αν εξετάσουμε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, εδώ στο σχετικό έγγραφο, στην τελευταία σελίδα, 12 στο αγγλικό κείμενο, υπάρχει ένα γράφημα σε ό,τι αφορά τις ε, τελικές συστάσεις. Και εκεί αναφέρονται μία-δύο στην εκπροσώπηση των ε, περιφερειακών αρχών και τοπικών αρχών ε, στην όλη διαδικασία και πώς, για παράδειγμα, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τρόπο έτσι ώστε να τροφοδοτούν ε, πληροφορίες, για παράδειγμα στην Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και σε άλλα θεσμικά οργανά της Ένωσης. Και αναφέρεται εδώ για παράδειγμα η δημιουργία περιφερειακών hubs, κέντρων δηλαδή, για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν την βελτίωση της νομοθεσίας, και εδώ δεν χρειαζόμαστε μια τέτοια εκπροσώπηση. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας δεν χρειάζεται δηλαδή η εκπροσώπησή τους ε, και ειδικότερα των, αυτών δηλαδή των εκπροσώπων των τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, και επίσης δεν θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όσες οργανώσεις συμμετέχουν στο των περιφερειών εκπροσωπούν πράγματι σωστά τους, ε, τους ε, πολίτες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να διασφαλίζουμε κάποιον τρόπο ότι πράγματι λαμβάνεται υπόψη η θέση όλων στο πλαίσιο της στήριξης αυτών των αξιών. Ένα δεύτερο ε, σχόλιο που θα ήθελα να κάνω έχει να κάνει με τη σελίδα 8 του κειμένου σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Εδώ στο σχετικό πλαίσιο αναφέρεται η αξιολόγηση πλήρω, στο ακέρο δηλαδή των δυνατοτήτων χρηματοδότηση των σχετικών οργανώσεων και τη εκπροσώπησή του. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε πάντοτε με τους ίδιους. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να περιληφθούν και εκείνοι οι οποίοι δεν γίνονται συνήθω ακούστε. Δεν έχουν δηλαδή, δεν ακούγεται δική του φωνή. Για παράδειγμα, διαφορετικές μειονότητες και ούτω καθεξής. Δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι εκπροσωπούνται και εκείνοι με κάποιο τρόπο. Επίσης, κατά τη δική μου άποψη, το κράτο ε, δικαίου ε, περιλαμβάνει και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την εφαρμογή του αυτού ακριβώς του κράτου δικαίου στην πράξη και νομίζω πως εδώ σε σχέση με αυτή την έκθεση που συντάσσεται ετησίω τίθεται και το ζήτημα του ε, ποιε είναι οι δυνατότητε πρόσβαση, ειδικότερα των γυναιτών στη δικαιοσύνη και ποια είναι τα εμπόδια για αυτήν την πρόσβαση. Εάν θέλουμε δηλαδή να ε, διασφαλίσουμε και τι ε, απαραίτητε αρχέ μα, δηλαδή η αρχή τη ισότητα των φύλων και το gender mainstream, η ένταξη δηλαδή αυτή τη διάσταση του φύλου στι βασικέ ε, ενωσιακέ πολιτικέ, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να μα αποσχολεί Και θα πρέπει, για παράδειγμα, να αυξήσουμε και το σχετικό προπολογισμό προ το ΆΕΓΕ, ούτω ώστε να αυξήσουμε και ε, τα σχετικά στατιστικά δεδομένα τα οποία παράγει, ειδικότερα διαχωρισμένα και αναφύλου. Με ανάλυση δηλαδή αναφύλου έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη ενημέρωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα τη διάσταση του φύλου σε ενωσιακό επίπεδο. Ευχαριστώ. η ε, ε, πάνελες να απαντήσω. Τώρα, πώ γίνεται αντιληπτή η εφαρμογή τη ενωσιακή νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Ναι, ε, έχουμε υπόψη μα πώ γίνεται αντιληπτή. Τώρα, αν είναι σωστή αυτή η αντίληψη, δεν έχει σημασία. Πάντω υπάρχει ότι ο νησιακό νόμο επιβάλλει νέε επιβαρύνσει. Η Επιτροπή Γιουνκερία έλεγε ότι θα είμαστε σημαντικοί για τα σημαντικά και ταπεινοί για τα δευτερεύουσα σημασία. Εμεί έχουμε τώρα αυτή την αρχή του ένα μπαίνει, ένα βγαίνει. Δηλαδή, θέλουμε να περιορίσουμε και να μειώσουμε, αν γίνεται, την γραφειοκρατία που δημιουργεί η εφαρμογή τη ουσιακή νομοθεσία επί των τελικών δικαιούχων. Βεβαίω, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία για του τελικού δικαιούχου η ενωσιακή νομοθεσία και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά. Και κάτι άλλο που επίση ισχύει είναι ότι πολλές φορές αυτά που παρουσιάζονται ως γραφειοκρατία, περιορισμοί επιβαρύνσεις δεν προέρχονται τελικά από το ενωσιακό δίκαιο. Στην ουσία δηλαδή κάποια κράτη-μέλη στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας το κάνουν ακόμη πιο ε, δυσχερές να εφαρμόσουν, την νομοθεσία, το λεγόμενο gold plating. Ορισμένες φορές τα κράτη-μέλη προσθέτουν γραφειοκρατία, προσθέτουν καθήκοντα και συνεχίζουν να λένε «Μα τα λέει η ενωσιακή νομοθεσία». Γι' αυτό υπήρξε το 2016 αυτή η διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθέτηση υπήρχε συγκεκριμένη ρήτρα για αυτό το gold plating και είπαμε στα κράτη-μέλη ότι όταν μεταφέρετε στο εθνικό δίκαιο την νομοθεσία να μην αξιοποιείτε την ευκαιρία για να προσθέσετε και δικές σας απαιτήσει. επιπλέον. Τώρα, τι εκπροσωπούν, ποιους εκπροσωπούν οι διάφορες διαβουλεύσεις και οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειών για παράδειγμα. Έχουμε ε, πολύ μεγάλη συνέστηση του θέματος αυτού. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία εκφράζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκλειστικά. Κατά τα άλλα κάνουμε διαβουλεύσεις με πολλού, αλλά ποτέ βέβαια δεν θα έχουμε την καλύτερη, την τέλεια εκπροσώπηση όλων των τμήματων της κοινωνίας, όλων των πολιτικών τάσεων, σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι περισσότερες απαντήσεις σε αυτές τις δημόσιες διαβουλεύσεις είχαν να κάνουν με την οδηγία για την θερινή ώρα. Λάβαμε 4,6 4,6 ε, απαντήσεις. Εκπροσω... Τι εκπροσωπούν. Όχι. Δεν εκπροσωπούν ε, τους πάντες. Διότι περίπου 3 εκατομμύρια ήταν ταυτόσιμες και προέρχονταν από ένα κράτος μέλος. Άρα, όταν εξετάζουμε το θέμα, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η γνώμη παντού στην Ένωση. Βεβαίω, ο τεράστιο αριθμό απαντήσεων που λάβαμε δείχνουν ότι υπάρχει θέμα ιδιαίτερα σε ένα κράτο μέλο το αντιλαμβάνονται ως θέμα περισσότερο από ό,τι στα άλλα αλλά για την Επιτροπή Περιφερειών δεν θεωρούμε ότι αυτά που μας δίνουν είναι η απόλυτη αντιπροσωπευτικότητα της εκπροσώπηση της κοινή γνώμης τώρα κοινωνία των πολιτών και ποιους χρηματοδοτούμε τώρα που θα έχουμε το νέο πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών στη νέα περίοδο της Επιτροπής πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερε δυνατότητε να χρηματοδοτήσουμε σωστότερα την κοινωνία των πολιτών. Και καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ ότι αν θέλουμε να υπάρξει νέου τύπου διάλογος για την κουλτούρα κράτους δικαίου, αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να συμπεριλάβει ε, μια πολύ ευρύτερη γκάμα από αυτούς που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στις συζητήσεις μας και τις διαβουλεύσεις μας και για την ε, ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αν δείτε τις πολιτικές κατευθύνες γραμμές της Προέδρου. Τονίζει ιδιαίτερα το κράτος δικαίου, την ισότητα των φύλων, πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε και τα δύο μαζί με μία προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και η Κάρεν. Αλλά σύντομα παρακαλώ Κάρεν, γιατί έχουμε και άλλο μελετή. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που δεν ήμουν στις παρουσιάσεις σας. Πολλοί συμμετέχουν στις δημόσιες ακροάσεις. Πολλοί ακούνε τις δημόσιες ακροάσεις και στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη γνώμη τους. Για παράδειγμα, μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων δεν έλαβε υπόψη η Επιτροπή τη γνώμη τους. Πώς θα αποφύγουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Γιατί βλέπουμε ότι στις ε, δημόσιες συζητήσεις συμμετέχουν όλο και περισσότεροι. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη τους και ότι το αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη τους. Μα φυσικά το λαμβάνουν υπόψη πολύ σοβαρά. όποιες απόψεις εκφράζονται κατά τις διαβουλεύσεις λαμβάνουν υπόψη σοβαρά. Κοιτάξτε, δεν κάνουμε μόνο διαβούλευση τώρα. Στην ε, εκτίμηση αντικτύπου έχουμε και μία συνόψη των απόψεων που εκφράστηκαν κατά την φάση διαβούλευσης και στα επεξηματικά μνημόνια ε, παρουσιάζουμε με σύντομο τρόπο την επίπτωση που είχαν αυτές οι γνώμες που εκφράστηκαν στην ε, διατύπωση της νομοθεσίας. Αλλά τι το θέμα εδώ, τι εκπροσωπούν αυτές οι απόψεις. Είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδυάσει για, και να καταλάβει τι εκπροσωπούν αυτές οι απόψεις τη συνοψίζουμε πάντα στα κείμενά μας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε όταν ε, κάνουμε την τελική διατύπωση της νομοθεσίας. Αλλά την τελευταία λέξη φυσικά την ε, έχουν οι συνομοθέτες. Εσείς και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Που απαντήσατε μερικές ε, πολύ δύσκολες ερωτήσεις από την Επιτροπή μας. και σίγουρα θα επανέλθουμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ και εσάς για τις ερωτήσεις σας. Η επόμενη παρουσίαση είναι η κυρία Ανδρέα Ρέντα, ο κύριος Ρέντα, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Υψηλού Ποπέδου, ο καθηγητής και δόκτωρ Ρέντα. Θα μας προσέξετε δύο εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί από την ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου, που έχουν να κάνουν με τι κρατικέ γραμμέ διοντολογία και τι ε, συστάσει για πολιτική και επενδύσει, πάντα για θέματα τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά βεβαίω θα τεθούν και ερωτήσει. Παρακαλώ κύριε Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ. περιμένω λίγο, γιατί βλέπω ότι κάποιοι έρχονται τώρα στην αίθουσα και κάποιοι φεύγουν. Και πάλι σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Λέγομαι Ανδρέα Ρέντα. Είμαι ένας από τους 52 που απαρτίζουν αυτή την ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη. Να σας πω πως συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα για την εντολή μας και για το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα για να επιτελέσουμε το έργο μας για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε την εντολή μας. Δε, θα σας τα πω ενδελεχώς όσον αφορά τα προβλήματα και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Πάντως, Όποιος θέλει μπορεί να μου υποβάλει ερωτήματα για να δούμε μαζί τα θέματα σε περισσότερο βάθος. Η εξέλιξη της προβληματικής για την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο ένωσης ανάγεται στο μακρότερο, μακρύτερο παρελθόν, απότερο παρελθόν τέλο πάντων, για όσον αφορά το πώς διαμορφώθηκε η πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και βέβαια άμεσα έχει εμπλακεί το γιατί υπάρχει για την ρομποτική, ένα ψήφισμα ε, και το αστικό δίκαιο. Ε, αυτό είναι, ήταν ένα πρώτο βήμα, ούτω ώστε επιγόντως να αναλυφθεί δράση για να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε τα προβλήματα, τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και προβλέπονται κάποια επιμέρους σημεία που αποτελούσαν μπούσολα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία την έκλεισε το Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να χάραξει ένα πλαίσιο πολιτικής για το θέμα μας και το Κοινοβούλιο. Ε, οργάνωσε μια σειρά συζητήσεων που ήδη βρίσκονται να εξελίξει. Πρώτα-πρώτα, κατά πόσο θα έχουν νομική προσωπικότητα τα FE αυτόνομα ρομπότ ή τέλος πάντων διάφορα ε, περίπλοκα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και όσον αφορά τη διακυβέρνηση επίσης και υπάρχει και η σχετική υπηρεσία ε, που θα μπορούσε να υπάρξει μάλλον για το κατά πόσον θα πρέπει επομένως μια τέτοια υπηρεσία να ιδρυθεί. Ακόμα ισχύουν ε, όλες αυτές οι συζητήσεις και μετά το πρώτο αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέλαβε τώρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγιναν μια σειρά πραγμάτων, δύο μόνο θα σα αναφέρω. Αλλά βέβαια το θέμα είναι πολύ ευρύτερο των όσων λέμε τώρα. Πρώτα-πρώτα έχουμε την συγκρότηση αυτή τη ομάδα φιλοπαίδου για την τεχνητή νοημοσύνη, που ο ρόλο του είναι να πάρει και συμβουλέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη γενικότερα. Είναι επομένω ανεξάρτητο σύμβουλο Οπότε πρώτα-πρώτα έχουμε την ανάπτυξη κάποιες διοντολογίες, κάποιες αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη και τα θέματα τα πιο λειτουργικά, δηλαδή τι γίνεται σε καθημερινή πρακτική, δηλαδή στην πράξη, δηλαδή τι κάνουν αυτοί που αναπτύσσουν την νοημοσύνη, αλλά και αυτοί που τη χρησιμοποιούν. Άλλο σημαντικό είναι κάποιες συστάσεις σε επίπεδο πολιτικής και όχι μόνο. Θα επανέλθω σε αυτό. Και άλλη πρωτοβουλία της Κομισιόν που σας ενδιαφέρει νομίζω είναι το ότι το ότι φτιάχτηκε αυτή η ευρεία μεγάλη πλατφόρμα που ήταν ένα βήμα για να συζητούνται τα πιο σημαντικά ζητήματα. Και αυτό λέγεται η Συμμαχία, ο Συνασπισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μια πλατφόρμα που ήλκησε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από του εμπλεκόμενου στο θέμα. Μιλάμε για 4.000 μέχρι σήμερα. Εκεί πέφτουν πολύ σημαντικέ πρωτότυπε ιδέες και ε, όλα αυτά βοηθούν και την ομάδα ψηλού επίπεδου του ειδικού. Και σε σχέση με αυτή την ομάδα να σας πω ακριβώς αυτό το, το πιο σημαντικό θέμα που φορά τη συζήτησή μας. Το ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες σε κάθε τομέα της τεχνητής ε, νοημοσύνης. Και αυτά έχουν σχέση με τις κατευθυντήριε της κυρίας Φόντερ Λάιν. Όσον αφορά τη διοντολογία, τα θέματα είναι σημαντικά για την Επιτροπή σας και ξεκινήσαμε με κάποια σχετικά απλή εντολή που κατέληξε να είναι πολύ πιο περίπλοκη. Δηλαδή να μπορέσουμε να επισημάνουμε τις βασικές αρχές που θα διέπουν την νοημοσύνη και να αντικατοπτρίζουν την κοινοτική προσέγγιση από την αρχή. Δηλαδή αυτό διέπνευσε τις εργασίες μας σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη για Ευρωπαίους σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Αρχές και στις συζητήσεις μας για το ποιες διοντολογικές αρχές θα είναι οι πιο δόκιμες στο πλαίσιο της Ένωσης ε, αμέσως αναδείχτηκαν και επισημάθηκαν προβλήματα, περιπλοκές, που όμως είναι απαραίτητε. Δηλαδή, το να παρεθμεί κανείς αρχές, κατά τη γνώμη μου, δεν λέει και πολλά για την ε, ομάδα μας, γιατί έχουμε ε, διάφορους φορείς, ιδιωτικού τομέα, κυβερνητικού τομέα, διάφορες ΜΚΟ. Ε, όλοι αυτοί ήδη έχουν επισημάνει αυτές τις βασικές αρχές. Και αυτοί που φτιάχνουν τα software παγκοσμίω ήδη έχουν λίστες με τέτοιες διοντολογικές αρχές. Δεν μας λείπουν τέτοιες αρχές που έχουν επισημανθεί. Ε, τα ίδια και τα ίδια. Διαφάνεια, ε, το να είναι κατανοητή η τεχνητή νοημοσύνη, να είναι ε, δίκαιη η διαδικασία, οι αλγόριθμοι, το πώς βρίσκονται οι αλγόριθμοι, να μην υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις, αυτό να είναι υποχρεωτικό. Ε, αυτά επαναλαμβάνονται συνεχώ από τους σχετικούς. Εμείς τα εξετάσαμε όλα αυτά και άρχισαμε να εκπονούμε με πρώτη δέσμη αρχών θεωρώντας ότι η Ευρώπη είναι διαφορετική. Δηλαδή, έχουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, έχουμε κάποιες βασικές αρχές και αξίες που ενσωματώνονται, θεμελιώνουν τις συνθήκες μας και την νομοθεσία μας. Οπότε η επαρρύθμιση απλώς των αρχών δεν λέει τίποτα, δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων του ότι θέλουμε να δούμε πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνολογία, σε σχέση με αυτές τις μη διαπραγματεύσιμες αρχές. Αυτή ήταν η πρώτη μας πρόκληση. Επομένω, πώς θα τα συναρμόσουμε αυτά, αυτές τις αρχές με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Με την ευρεία είναι. Και όχι με την έκφανσή τους στο κοινωτικό δίκαιο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα για προστασία των ανθρωπίνων και ομάδων κοινωνικών μέσω της ατομικής ηθικής. Πέραν δηλαδή της ιδιότητας του πολίτη. Τα λέω όλα αυτά, τώρα και επιτρέψτε μου να κάνω αυτές τις υπεραπλουστεύσεις. Άρα αυτό αποφάσισαμε ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει βασικά να εδράζονται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό που λέμε ηθική, τεχνητή νοημοσύνη. Α, αυτή δηλαδή που συμμορφώνεται με το δίκαιο. Με τον νόμο. Όπως ε, Ισχύει σήμερα και όπως θα δημορφωθεί στο μέλλον. Άρα, τελικά, δεν πρόκειται για ηθική τέχνη νομοσύνη, αλλά για αξιόπιστη. Άρα αυτό είναι, συμμόρφωση ηθική. Επομένως, πέραν αυτών, πέραν αυτής της συμμόρφωσης που επιβάλλεται, επίσης επισημάναμε μια σειρά ηθικών αρχών, ίσως να τις ονομάσουμε αρχές πέραν της συμμόρφωσης. ηθική πέραν τη συμμόρφωση. Δηλαδή, αφού κανεί συμμορφώνεται με τον νόμο, πώ κανεί θα προσανατολίσει αυτήν την ε, τεχνητή νομοσύνη, ώστε να είναι αξιόπιστη. Και άρα αυτό είναι ο άλλο πυλώνα μα, δηλαδή να επισημάνουμε όλε αυτέ τι ηθικέ αρχέ, τι ονομάζουμε αυτέ τι τέσσερι αρχέ που είναι οι κατευθυντήριε ε, γραμμές μας, οι οποίε προβλέπονται για να προσανατολίζουν, να καθοδηγούν την ανάπτυξη τη τεχνητή νοημοσύνη προ αυτό που θεωρούμε ότι είναι η προϋπόθεση για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στην τεχνολογία από τον κόσμο, από τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, από τα θεσμικά όργανα. Οπότε, θα επανέλθουμε σε αυτό για να συμπληρωθεί αυτό το μοσαϊκό. Γιατί έχουμε και τον τρίτο πυλώνα για να μπορέσουμε να είμαστε αξιόπιστοι και εμείς θεωρούμε ως ομάδα ότι χρειάζεται να υπάρχουν προϋποθέσεις για περισσότερη εμπιστοσύνη. Μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα, Oxford Analytica και ένα σωρό άλλα, όλα όσα έχουν γίνει και οδήγησαν σε αυτή την ε, μείωση της εμπιστοσύνη για τις πλατφόρμες και λοιπά για την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα τώρα έχουμε αυτό το πλαίσιο για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε και αυτό το τρίτο πυλώνα που ονομάζεται το κοινωνικό τεχνικό στεγανό της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα Μιλάμε για το πώς θα είμαστε πιο ανθεκτικοί σε κυβερνοεπιθέσεις, να μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργικότητα, μακροπρόθεσμα. Όλοι όσοι αναπτύσσουν την νοημοσύνη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ισχύουν όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Και όλοι οι κίνδυνοι της λειτουργίας έχουν καλυφθεί και δεν υπάρχει περιθώριο. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να ισχύει 100% ε, και αυτό να ισχύει συνεχώ κάθε λεπτό γιατί τα πράγματα εδώ είναι πολύ περίπλοκα αλλά τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα να έχουμε τελευταία λέξη τεχνολογία. να εξασφαλίσουμε ότι όχι μόνο ισχύουν οι προποθέσει για τη θωράξη αλλά και ότι θα υπάρχουν κάποια αμυντικά μέτρα τα οποία να ενεργοποιούνται όταν κάτι συμβεί να, η διακυβέρνηση από πλευρά ασφάλεια και αξιοπιστία. άρα αυτό που λέγαμε στην αρχή η ηθική η Έγινε τώρα έτσι με αυτούς τους τρεις πυλώνες συμμόρφωση, ε, στεγανότητα, ηθικότητα. Οπότε, σε αυτό το την ευθυγράμμιση των, των αρχών, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι πάμε ακόμα πιο βαθιά στις κατευθυντήριες που δημοσιοποιούμε στις 9 Τετάρτου φέτος. Γιατί τότε είναι η μέρα της ψηφιακής τεχνολογίας και εκεί απαριθμούμε Εκεί εντοπίζουμε αυτές τις ηθικές αρχές και τις μετατρέπουμε, τις, τις, εξελίσσουμε σε επτά προϋποθέσεις. Να, το νέο στοιχείο που ίσως μια μέρα, μια μέρα μπορεί να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Πλαίσιο πολιτικής. Ήταν η πρώτη απόπειρα αυτές οι προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε μια λίστα αξιολόγησης. Στην αρχή λέγαμε ότι αυτό θα ήταν αυτοαξιολόγηση. Δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά να τα χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν το ότι αν όσα κάνουν οδηγούν στο, στο αξιόπιστον κλπ. κλπ. Αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό που προτείναμε, αυτού του είδου η λίστα, είναι αυτοαξιολόγηση. 131 άρθρα Φυσικά και είναι μακροσκελής, το ξέρουμε. Αλλά είναι η πρώτη απόπειρα να πάμε παραπέρα από αυτό που τόσα χρόνια ήταν η απαρίθμηση ειδικών αρχών που δεν είχαν κανένα συγκεκριμένο χαρακτήρα που να επιδέχεται η υλοποίηση. Να κάνουμε μερικά βήματα παραπάνω από την ανάπτυξη για να δώσουμε κάποιε ενδείξει σε αυτούς που χρησιμοποιούν, που εμπλέκονται, που έχουν σχέση τέλο πάντων με την ε, ε, τάφνη. Οπότε όλα αυτά να εξασφαλίσουν το ότι η διαδικασία της ανάπτυξης και η περισάρκωση αυτού του συστήματος ε, της διάχυσης θα διέπεται από όλες αυτές τις λίδες ασφαλείας. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Α, γιατί φτάσαμε σήμερα στη μέση παρουσίαση. Το κατάλογο αυτό τον εκπονήσαμε σε πολύ διαφορετικό κλίμα το οποίο νέο κλίμα διαπίστωσε σε μια χθεσινή συνεδρίαση. Τα εργαλεία αυτά τα εκπονήσαμε όταν η DG Connect της Επιτροπής μας έλεγε ότι προς το παρόν θα προτιμούσαμε την αυτορύθμιση ως ε, πιο επιθυμητή λύση. Και είχαμε μια πολύ πιο ε, στάση αναμονής για να δούμε αν ε, τελικά θα υπήρχε ε, αυθόρμητη συμμόρφωση με τις αρχές. Εάν έτσι δηλαδή ο κλάδος θα εφήρμοζε αυτές τις αρχές αυθόρμητα, χωρίς να χρειαστεί ε, η παρέμβαση της πολιτικής. Η κατάσταση όμως σήμερα έχει αλλάξει πολύ. Η πρόεδρος Φοντερ Λάιν ανακοίνωσε ότι εντός των πρώτων 100 ημερών τη θητείας τη, όποτε και να αρχίσουν, θα υπάρξει πρωτοβουλία για τις ε, επιδράσεις στον άνθρωπο και στην κοινωνία τη τεχνητής νοημοσύνης. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι καθεντήρες γραμμές δεοντολογίας μας θα είναι τμήμα αυτή τη πρωτοβουλία. Όταν παρουσιάσαμε λοιπόν αυτές τις, αυτές τις καθευτήριες γραμμές για, για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, θεωρούσαμε ότι κάναμε το πρώτο βήμα μιας μεγάλης διαδικασίας. Και μετά είχαμε διάφορες πολιτικές δράσεις με ερευνητικού οργανισμούς στην κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσει, θεσμούς. Για να δούμε εάν αυτός ο κατάλογος αξιολόγηση που ξέρουμε ότι είναι ακόμη πρόχειρος, πόρο απέχει από την τελική του έκφανση, θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο κατάλογο να εκλεπτυνθεί για συγκεκριμένους ε, κλάδους, συγκεκριμένες χρήσεις, ακόμη και αν είναι δυνατόν για συγκεκριμένες εταιρείε. Ανάλογα με τους κινδύνους που δημιουργούνται από το βαθμό χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Κάναμε λοιπόν μία έρευνα μεγάλης ε, διάστασης Συλλέγουμε ήδη τα στοιχεία που μπορούν να μας τα στείλουν πάνω μέχρι το τέλος του μήνα. Ελπίζουμε να λάβουμε μερικές εκατοντάδες απαντήσεις για να κάνουμε μια αποτίμηση. Σε τι βαθμό ο κατάλογος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα, εάν γίνεται εύκολα κατανοητός και εάν δημιουργεί διοικητικό βάρος μεγάλο για όσους θέλουν να τον εφαρμόσουν. Και αν κάποιες εταιρείες ή η τεχνική της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν ήδη να βασιστούν στις διαδικασίες που προβλέπει, όπως και οι διαδικασίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων, εάν μπορούν να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Σε ένα βαθμό βέβαια θα μειωθεί το επιπλέον άχθος ε, εφόσον ήδη κάποιες ε, προϋποθέσεις προβλέπονται ήδη από άλλα νομοθετήματα. Επίσης, Υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που λέγεται Τεχνητή Νοημοσύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω αυτού κάναμε 50 συνεντεύξεις με διάφορες εταιρείε από διάφορες χώρες, διαφόρων τύπων, διαφορετικού μεγέθους, ακόμη και με μονομένους ερευνητέ και με δημόσιους οργανισμούς, για να βρούμε εάν αυτός ο κατάλογος είναι τελικά εύχριστος και πώς πρέπει να τον αναθεωρήσουμε. Επίση είπαμε στη Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη να μας πει πολύ πιο ειλικρινά τι απόψεις τη. Θέλουμε κάθε σχόλιο. Τις απαντήσεις αυτές θα τι έχουμε μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Έμαθα χθε. Θα αρχίσουμε να αναθεωρούμε από τι 16 Δεκεμβρίου αυτό το κατάλογο κριτηρίων για να καταλήξουμε σε ένα πιο εύχριστο αποτέλεσμα που θα είναι το πρώτο τέτοιου τύπου στην ε, χρήση της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Κανένα, καμία άλλη χώρα, ε, κανένας άλλος τομέας χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Θα, είμαστε λοιπόν, έστω για να κάνουμε λάθη, πρωτοπόροι, αν τελικά εγκρίνουμε, αν τα όργανα της Ένωσης εγκρίνουν αυτό το κατάλογο. Κοιτάξτε, μπορεί Αυτά που σας λέω βέβαια να είναι απλώς ε, οι δικέ μου φαντασιώσεις. Δεν ξέρουμε. Ας πει κάποιος, αν μας πει κάποιος ότι αυτός ο κατάλογος εταιρείων θα μπορούσε να είναι τμήμα μιας διαδικασίας πιστοποίησης. Δηλαδή οι εταιρείε δεν θα πρέπει απλώς να επιδιώκουν να λειτουργούν με αυτήν την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να απαιτείται να εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια. Οπότε αυτός ο κατάλογος θα πρέπει να μεταφραστεί σε κάτι που να μπορεί να αξιολογηθεί και ποσοτικά, να μπορεί να βάλεις βαθμό. Για παράδειγμα, για τις διακρίσεις, για το σεβασμό για την ε, αυτονομία των ατόμων. Να λέμε ότι ο τάδε οργανισμός λαμβάνει επαρκή μέτρα, ούτω ώστε το προϊόν του να θεωρείται αξιόπιστο και να πάρει τον τάδε καλό βαθμό. Και να υπάρχει και βάση. Να δούμε αν είναι κάτω από τη βάση. Να επανέλθω βεβαίω από αυτού, να σε ενημερώσω, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουμε λάβει τα στοιχεία. Όταν και εμεί λοιπόν θα ξέρουμε περισσότερα. Για να δούμε δηλαδή και πόσο φιλόδοξε θα είναι οι προτάσει τη Επιτροπή που θα, που θα διατυπωθούν ε, προσεχώ. Έχω ασχοληθεί πολύ και με την καλύτερη νομοθέτηση ω πανεπιστημιακό. Ξέρω ότι αν υπάρξει μια πρωτοβουλία τι 100 πρώτε μέρο και μετά θα δούμε αυτήν την ε, ε, αρχική εκτίμηση αντικτύπου. Μετά θα γίνει διαβούλευση με βάση αυτήν την αρχική εκτίμηση αντικτύπου. Έτσι είναι η διαδικασία μας. Όλα αυτά θα γίνουν πριν λάβετε την πρόταση. Έτσι θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Γιατί αυτή η προπαρασκευαστική διαδικασία που είναι τμήμα του θεματολογίου της καλύτερης νομοθέτησης θα απασχολήσει πολύ τις υπηρεσίες τις πρώτε 100 μέρε. Περιμένω η Κομισιόν να ξεκινήσει, αλλά αμέσω μετά θα δούμε τις πρώτες προτάσεις που θα υποβληθούν. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα. Και αν έχετε ερωτήσεις ε, για αυτόν τον κατάλογο, ευχαριστώ. Δεν θα αναθεωρήσουμε όμως ε, τις κατευθυντήριε γενικά, αλλά μόνο αυτό το κατάλογο. Αυτό μπορεί να γίνει αργότερα. Αυτή η ιδέα αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη είναι ε, και ένα τμήμα ε, του δεύτερου κλάδου δραστηριότητας που έχουμε αναλάβει. Είναι οι συστάσεις για την πολιτική και τις επενδύσεις. Στις 26 Ιουνίου τρέχοντος υποβάλαμε ένα έγγραφο. Είναι αρκετά ευρύ, συστημικό θα έλεγα οικοσυστημικό αν θέλετε για την τεχνητή νοημοσύνη για να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για αυτή την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη και να βεβαιωθούμε ότι έχουν συνέστηση οι νομοθέτες ότι πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη αυτά παντού. Δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα αν δεν είναι ισχυροί οι θεσμοί, αν δεν υπάρχει ένας δημόσιος τομέας που να δρά ως καταλήτης. Δεν θα υπάρξει ισχυρή, ισχυρό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης αν δεν υπάρξει επαρκής συνειδητοποίηση από πλευρά τη κοινωνία των πολιτών και αν δεν υπάρξουν ε, επαρκή, αρκετά μάλλον άτομα με επαρκεί δεξιότητε για να την εφαρμόσουν. Και χρειάζεται επίση έρευνα και καινοτομία. Και κανόνε που να βοηθούν τη μόνιμη καινοτομία συνεχώς με πλήρη σεβασμό των αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ήδη ανέφερα. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια σειρά από πολλε ειναι είναι. Μια-δυο θα αναφέρω για να σας δώσω μια ιδέα. Πώς λειτουργεί το σύστημα. Το πιο σημαντικό τμήμα, νομίζω, των συστάσεων, δεν ξέρω, κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να διαφωνούν, γιατί ο καθένα μας ασχολείται με διαφορετικά θέματα. Αλλά νομίζω ότι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή σα είναι ότι προτείνουμε ένα σύστημα που να βασίζεται στη διαχείριση κινδύνου δεν ζητάμε από κάθε τεχνικό τεχνητής νοημοσύνης να έχει το ίδιο επίπεδο μέτρων αντιμετώπισης των ε, κινδύνων. Γιατί οι διαφορετικές εφαρμογές ε, της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν διαφορετικού τύπου και επίπεδου κινδύνους. Και όσοι πρόκειται να δημιουργήσουν τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης αλλά κύριοι, ιδιαίτερα λοιπόν αυτοί οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα πρέπει να εκτιμούν τον κίνδυνο που θα δημιουργήσει το προϊόν τους και να εγκρίνουν και τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπιση του κινδύνου. Ένα σύστημα που βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου με τα αναλογικά μέτρα, δηλαδή αναλογικά προς τον κίνδυνο, δεν θέλουμε όμως το σύστημα αυτό να είναι υπερβολικά προληπτικό υπερβολικά επιφυλακτικό. Ξέρουμε ότι η αρχή της πρόληψης είναι σημαντική. Αλλά εάν ε, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο ενός προϊόντος τεχνητής νοημοσύνης και ο κίνδυνος από το να πάει στραβά ένα σύστημα ε, θα έχει, να έχει τεράστιες επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλου, τότε βεβαίως θα υιοθετήσουμε την αρχή της πρόληψης. Γι' αυτό προτείνουμε ένα τέτοιο σύστημα. Και το σημαντικό είναι ακριβώς αυτό, ότι αυτοί που αναπτύσσουν και μετά εφαρμόζουν τα προϊόντα τεχνητή νοημοσύνης είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του κινδύνου. Ξέρετε, τόσο περισσότερο διαδίδονται αυτά τα προϊόντα στην κοινωνία ούτω ώστε ε, όχι μόνο τα άτομα να αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη να επιδρά με την τεχνητή νοημοσύνη και να παράγουν στοιχεία όλα αυτά, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε σε καταστάσει όπου ένα σύστημα που μπορεί να λειτουργεί πολύ σωστά, που έχει ελεγχθεί σωστά σε ένα ε, ερευνητικό περιβάλλον, μπορεί να ξεφύγει εντελώ τη στιγμή που θα αρχίσει στην κοινωνία, γενικά στον πραγματικό κόσμο, να αλληλεπιδρά με άλλου αλγορίθμου. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ καλή εξάντια αξιολόγηση, αλλά ένα πλήρη κύκλο αξιολόγηση για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί και πολλά, πολύ τέτοια προϊόντα να διασφαλίσει ότι οι τελικοί χρήστε, η οικονομία, το περιβάλλον δεν θα κινδυνεύσουν. Πρέπει να γίνονται διαρκώ έλεγχοι και αν προκύπτουν προβλήματα λαμβάνονται μέτρα. Ακόμη και μετά την πώληση ενό συστήματο από του πολιτέ για να διατηρηθεί η αξιοπιστία του. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ περίπλοκα. Αλλά είναι μια εξέλιξη. Είναι απλώς μια εξέλιξη προϊόντων που ήδη υπάρχουν. Και βεβαίως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ε, είναι κάπως απρόβλεπτα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κάτι άλλο. Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα που πάντα αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πολιτική να παρακολουθεί τους ρυθμούς εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλάζουν συνεχώς τα προβλήματα και οι κίνδυνοι. Οι νομοθέτε, όχι μόνο σε εσά, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παντού οι νομοθέτες, λαχανιάζουν για να προλάβουν την ε, ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ε, κάνετε την νομοθεσία σας. Πρέπει λοιπόν βεβαίως πάντα να βασίζεστε σε αρχές, να βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά να είστε ταχεί και ευέλικτοι. Η εξέλιξη, για παράδειγμα, των ε, ρυθμιστικών λύσεων. Να ελέγχουμε κάποιες λύσεις ε, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο πριν τις περάσουμε στην αγορά. Όλα αυτά πρέπει να είναι αρχές της πολιτικής της Ένωσης. Γιατί αυτό που διαπιστώνουμε στην εργασία μας είναι ότι όχι μόνο εσείς ως ενωσιακοί νομοθέτες. Ούτε καν οι οργανισμοί τυποποίησης δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το ρυθμό εξέλιξης ε, των λεγόμενων βαθέων ψευδών. Κάθε δύο εβδομάδες, το λεγόμενα deep fakes, κάθε δύο εβδομάδες αλλάζει η κατάστασή τους. τη στιγμή που δημοσιεύονται βιβλία για αυτά τα θέματα, ένα χρόνο μετά δηλαδή την ε, ε, εμφάνιση ενός φαινομένου είναι ήδη ξεπερασμένα. Έχουμε δημοσιεύσει αυτές τις ε, συστάσεις και αν έχετε ερωτήσεις να τις ακούσω. Τέλος. Όχι μόνο ε, βρισκόμαστε στη φάση της εκπόνησης των κατευθυντήρων γραμμών και της αξιολόγηση τους, αλλά η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου έχει την εντολή μέχρι τα μέλη του 2020 να κάνει το εξής να οργανώσει μια σειρά από θεματικά workshop έτσι ώστε σε αυτές οι συστάσεις να εξατομικευτούν, αν θέλετε, να γίνουν πιο συγκεκριμένες σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους επιμέρους τομείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είμαστε και επιλεκτικοί εδώ, γιατί δεν έχουμε και απεριόριστους πόρους στη διάθεσή μας. Άρα λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από streams, ροές δηλαδή εργασίας, σε ό,τι αφορά τρεις βασικά αρχικούς κλάδους, τους οποίους έχουμε εντοπίσει και στους οποίους θέλουμε πραγματικά να έρθουμε σε επαφή με τους stakeholders έτσι ώστε οι συστάσεις μας να είναι πιο εξειδικευμένες για τον κάθε σε κλάδο. Καταρχήν έχουμε να κάνουμε με τον δημόσιο τομέα, τις δημόσιες υπηρεσίες, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά μια επίσημη αναγνώριση στο πλαίσιο των τελωνίων ή δημόσιοι χώροι και γενικά διάφορες τομεί μέσα στο δημόσιο τομέα. Δεύτερο τώρα κλάδο, δεύτερο τομέα στον οποίο εστιάζουμε είναι αυτό τη μεταποίηση. Και αυτό και ειδικότερα δηλαδή σε ό,τι αφορά τις εφαρμογε b B2B από επιχειρήσει προς επιχειρήσει και την τεχνητή νοημοσύνη, θεωρούμε πως εδώ πολλά μπορεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση σε ό,τι αφορά και την ανταγωνιστικότητα και ειδικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα τρίτο τομέα είναι αυτός ε, της ε, υγείας γιατί εδώ έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και μεθοδολογικά και διαδικαστικά σε ό,τι αφορά δηλαδή την χρήση, την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά και ακριβώ επειδή έχουμε και γρήγορε εξελίξει σε αυτού του τομεί. Άρα λοιπόν αυτοί είναι τρει τομεί ε, του οποίου θα εξετάσουμε. Επίση θα υπάρξουν και κάποια streams σε ό,τι αφορά τι οικονομικέ υπηρεσίε και τον τομέα τη γεωργία, αλλά χωρί δηλαδή επίσημη εποπτεία από την πλευρά τη ομάδα πυρογνωμών υψηλού επίπεδου. Δηλαδή το κάνουμε πιο εξατομικευμένα, εγώ ε, ειδικό και ούτω καθεξή. Από εκεί και μετά έχουμε και μια ιδιαίτερη εστίαση στην κυβερνοασφάλεια ε, καθώς μας απασχολεί ιδιαίτερα και το σύστημα πιστοποίησης το οποίο έχει αρχίσει να ε, δημιουργείται τώρα στο πλαίσιο ακριβώς της ε, κυβερνοασφάλειας. Μία τελευταία δήλωση θα ήθελα να κάνω. Όλα αυτά είναι σημαντικά όχι επειδή η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ασήμαντη. Αλλά αν μου πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτύχει τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030 χωρίς την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθώ εγώ να πω και στο πλαίσιο της ε, ε, ομάδας για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το ε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Αντίστροφη είναι ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την Ευρώπη. Ειδικότερα δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με το Internet of Things μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα τη προσπάθεια σε ό,τι αφορά ε, την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και την αύξηση τη ανταγωνιστικότητά μα. Και είμαι στη διάθεσή σα βέβαια για ερωτήματα. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι αυτό ο τομέα δεν είναι αμυγό, αν θέλετε, στι αρμοδιότητε τη ε, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αλλά συνήθω τα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη δεοντολογία έχουν να κάνουν ακριβώ με τι προκλήσει που αντιμετωπίσουμε και προσπαθούμε εδώ λοιπόν, να εμβαθύνουμε την κατανόησή μα για αυτά τα ζητήματα. Αυτά λοιπόν από την πλευρά μου και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο, ε, για αυτήν την πολύ διεξοδική παρουσίαση. Επειδή έχουμε πολλού ομιλητέ, Τζάκι Τζόν, και Justin Bieber είναι οι τρει πρώτοι ομιλητέ που θα πάρουν το λόγο και στη συνέχεια επόμενο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Τζάκι Τζόν. Ε, ακούσαμε πάρα πολλά. Οπότε θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξή. Μα είπατε ότι εσά σα απασχολεί το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή την αποφυγή των διακρίσεων, μία, ένα από τα βασικά κριτήρια ακριβώ είναι αξιοπιστία. Δηλαδή να λαμβάνετε υπόψη επικοινωνία, να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση, να μην υπάρχουν δυσμενεί διακρίσει. Σα ρωτώ λοιπόν πώ ακριβώ αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη. Πώ μπορείτε δηλαδή να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίο, για παράδειγμα, θα αποφεύγει ακριβώ την επιβολή διακρίσεω βάρο των γυναικών. Ευχαριστώ. Λέει πρόεδρο, παρακαλώ, Μέρκελ. Ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εκείνο που μου άρεσε ήταν το γεγονός ότι δεν δόθηκαν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, λύσεις τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Εκείνο που θα ήθελα να ακούσω εγώ είναι λίγε περισσότερε ε, λεπτομέρειε σε σχέση με αυτό το κατάλογο αξιολόγηση, το assessment list. Γιατί πολλά από τα ζητήματα που αφορούν ε, την τεχνητή νοημοσύνη έχουν να κάνουν με το πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη λογοδοσία, το accountability, πώ μπορούμε να ε, διασφαλίσουμε ταυτόχρονα το ποικιλόμορφο χαρακτήρα έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή να λαμβάνει υπόψη όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και όχι μόνο μερικές από αυτές. Και επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω να αναφερθείτε στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτελέσει σιγά σιγά έναν γενικό όρο που περιλαμβάνει όλες τις νέες τεχνολογίες τις οποίες ε, δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς πώς λειτουργούν. Δηλαδή πώς η δική σας ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου ορίζει επακριβώς την τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη έμφαση που δίνετε στο ζήτημα της αξιοπιστίας. Ευχαριστώ. Λέει πρώτος ο κύριος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την παρουσίαση. Τρία ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Καταρχήν, η Επιτροπή μα είπε πω θέλει να αξιοποιήσει τι συστάσει αυτή τη ομάδα εμπειρογνωμόνων ω βάση για την πρόταση μια νομοθεσία. Παρότι βέβαια η εν λόγω οι συστάσει δεν είχαν αυτόν τον στόχο. Οπότε θα ήθελα να σα ζητήσω να σχολιάσετε την κριτική που ασκήθηκε ε, απέναντι σε αυτή την ομάδα ε, εμπειρογνωμόνων ότι δηλαδή υπερεκπροσωπείται από τον βιομηχανικό κλάδο, γιατί αντιθέτω δεν υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση από την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Πράγματι λοιπόν αυτέ οι συστάσει θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ω βάση για την διατύπωση νομοθεσία. Επίση, θα θέλατε για παράδειγμα να λάβετε υπόψη σα άλλε συστάσει, για παράδειγμα όπω αυτέ τη Επιτροπή Διοντολογία τη ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία. Ε, δεύτερο ερώτημα. Όταν κάνουμε ε, λόγο για τεχνητή νοημοσύνη και την σχετική ε, δεοντολογία ηθική, ποιοι αλγόριθμοι θεωρείτε πω είναι ανήθικοι, α το πούμε έτσι, που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια παραδείγματα και δεν άκουσα να αναφέρετε κάτι τέτοιο. Και τρίτο ερώτημα. Ε, ποια δικαιώματα θα πρέπει να έχουν οι πολίτε εκείνοι για του οποίου ενδεχομένω να υπάρχουν αρνητικέ συνέπειε, εφόσον για παράδειγμα υπάρξει κάτι, μια απόφαση βάρο του, στην οποία θέλουν να προσβάλλουν. Πώς, ποια, ποια μέσα προσφυγή, αν θέλετε, θα έχουν απέναντι σε κάτι τέτοιο. Αν για παράδειγμα υποστούν δυσμενή διάκριση, τι είδου δικαιώματα λοιπόν θα πρέπει να είναι διασφαλισμένα για αυτού του πολίτε. Ευχαριστώ, λέει ο Να ακούσουμε Και μετά θα ακούσουμε και άλλου συναδέλφου. Ναι. Ε, Απαντώντα πολύ σύντομα στο ερώτημα του τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για την ε, Ευρώπη. αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα αποτελεί ουσιαστικά το προϊόν της ε, τεράστιας ε, διαθεσιμότητας ε, δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας. Δηλαδή, κατά τις πρώτες του δεκαετίες το διαδίκτυο ή το World Wide Web, για να το πούμε πιο σωστά, οδήγησαν σε μια τεράστια διαθεσιμότητα δεδομένων, μεγάλο όγκο δηλαδή δεδομένων, ειδικότερα προσωπικών δεδομένων που παράγονται από του χρήστε. Και αυτό δημιούργησε με τη σειρά του ανάγκη σε επίπεδο έρευνα σε ό,τι αφορά τύπου τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι ακριβώ ε, είναι ιδιαίτερα ε, χρησιμοποιούν μεγάλο όγκο τέτοιων δεδομένων. Γι' αυτό συχνά πράγματι γίνεται λόγος για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που εννοούμε είναι το machine learning, δηλαδή εκμάθηση, αν θέλετε, από υπολογιστικέ μηχανέ που αποτελεί κάτι πολύ συγκεκριμένο και ακριβώ είναι. Ε, απαιτεί πολύ μεγάλο όγκο ε, δεδομένων. Άρα λοιπόν κινούμαστε, ε, αρχίζουμε να απομακρυνόμαστε από συστήματα τα οποία ακολουθούν πολύ συγκεκριμένου ε, κανόνε, όπω για παράδειγμα οι που χρησιμοποιούμε σήμερα, που τροφοδοτούνται δηλαδή με δεδομένα, κάνουν υπολογισμού και παρέχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και κινούμαστε όλο ένα και περισσότερο προ ε, μηχανήματα τα οποία ουσιαστικά ε, μέσω δικών του συστημάτων ενευρών, κάνουν τους δικούς υπολογισμούς και, τους, και ζητείτε να επαληθευτεί κατά πόσο τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν είναι σωστά ή όχι. Ε, για να γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο, ε, χρειάζεται τεράστιο όγκο δεδομένου και αποτελεί προσωμείωση, αν θέλετε, κάποια ευφυία, αλλά δεν αποτελεί ευφυία πραγματικά intelligence. Αποτελεί προσωμείωση ευφυία και αφορά σε πολύ συγκεκριμένα, σε πολύ συγκεκριμένε πράξει, τι οποίε δηλαδή επιτελούν τέτοιου είδου συστήματα. Γιατί συχνά τίθεται και αυτά τα ερωτήματα σε ό,τι αφορά αυτή την ευθεία. Ε, συχνά λοιπόν βλέπουμε να, έχουμε, να έχουν διάφορε χώρε τεράστιο όγκο δεδομένων, ειδικότερα ε, σε ό,τι αφορά το machine learning, αυτό το τομέα, ε, σε σχέση με εφαρμογέ, για παράδειγμα, από επιχειρήσει προ ε, τελικού πελάτε. Όπω για παράδειγμα στην περίπτωση του Netflix ή στην περίπτωση του Google. Τέτοιου είδου λοιπόν εφαρμογέ, οι οποίε για να λειτουργήσουν χρειάζονται πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Και όσο μεγαλύτερο ε, είναι αυτό ο όγκο δεδομένων, τόσο πιο ακριβή είναι αυτά τα συστήματα και πιο αποτελεσματικά. Χωρί αυτό να σημαίνει βέβαια ότι κάτι τέτοιο είναι πάντοτε επιθυμητό. Υπάρχει λοιπόν η τάση σε σχέση με αυτού του είδου τι εφαρμογέ να ε, υπάρχει ε, μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στην ακρίβεια αφενό και, την, το, το, το, το, να είναι επεξηγήσιμη μια τεχνολογία αφετέρου. Ε, δηλαδή, Εάν, για παράδειγμα, εφαρμόσουμε μια τέτοια τεχνολογία, ούτω ώστε να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση ενό ε, συγκεκριμένου συστήματο δεδομένων, δεν χρειάζεται να είναι επεξηγήσουμε αυτό το δεδομένο. Αλλά αντιθέτω, όταν έχουμε ένα σύστημα διαχείριση ε, δεδομένων, χωρίς, ε, και για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο χωρί να μπορούμε να εξηγήσουμε το γιατί γίνεται αυτό, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό το αναφέρω σε σχέση με δύο περιπτώσεις που προέκυψαν στις Ηνωμένες σε σχέση δηλαδή με ε, ε, πράξεις και ακριβώς την μη πρόσβαση σε τέτοιου είδους ε, δεδομένα, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα επεξήγηση του γιατί ακριβώς αυτό είχε προβλεφθεί. Και αυτό σε επίπεδο του οικονομικού δικαίου των, της, των ΗΠΑ. Ακριβώς αυτό δηλαδή καταδεικνύει τον προβληματισμό που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους ε, συστημάτων. Και εδώ δεν αναφέρομαι για παράδειγμα σε ε, σε ζητήματα αποκλειστικά και μόνο προσωπικών δεδομένων, γιατί σε εκείνε τι περιπτώσει πάντοτε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τέτοιου δεδομένων θα πρέπει να είναι δυνατόν να δοθεί μια εξήγηση. Γιατί πάντω αναφέρθηκα σε αυτό το ζήτημα, Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο αυτό το machine learning. Υπάρχει και ένα άλλο νέο κύμα τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο δεν απαιτεί τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων και ενδεχομένω θα είναι πιο χρήσιμο σε ό,τι αφορά ακριβώ ε, και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την ανταγωνιστικότητα τη Ένωση. Και σε τι αναφέρομαι εδώ, σε εφαρμογέ B2B, από επιχειρήσει προ επιχειρήσει, στι περισσότερε περιπτώσει. Και τώρα οι επιχειρήσει και οι πυρογνώμονε εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα όλο και είναι πιο εγκύτερα στα ίδια τα things, τα πράγματα δηλαδή, στα οποία αναφέρονται, χωρί να είναι ανάγκη δηλαδή να υπάρχει συγκέντρωση όλων αυτών του, του μεγάλου όγκου δεδομένων. Δηλαδή, αυτά γίνονται μέσω ακριβώ των διαπαφών που έχουμε με, τα διάφορα, με διάφορε συσκευέ, τα διάφορα μηχανήματα, τα εν λόγω συστήματα. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα χρειάζεται πια αυτό τεράστιο όγκο δεδομένων όπω το προηγούμενο κείμενο. Θα έχουμε μικρά δεδομένα, small data όπω λέγονται. Αυτά θα μα επιτρέψουν να φέρουμε μια επανάσταση στη Γεωργία, να ε, ε, εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία μας, να βελτιώσουμε την δημόσια υγεία μας. Ε, γιατί είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μα ενδιαφέρει εδώ δηλαδή να βελτιώσουμε την τεχνολογία, να μπορούμε να βγάζουμε καλύτερε σέλφι. Όχι, θέλουμε συστήματα ακριβώ τα οποία θα βελτιώσουν την, το βιομηχανικό μα κλάδο, τη γεωργία μα και ούτω καθεξή. Αλλά αυτά τα συστήματα ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί. Όταν λοιπόν θα καταρτήσετε την νομοθεσία σα και θα δημιουργήσετε τα προαπαιτούμενα για την ε, σχετική τεχνολογία που θα αξιοποιούν οι δημόσιε αρχέ, εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ακριβώ να προβλέψετε τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία θα είναι δυνατόν χρησιμοποιούνται, ώστε να μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει, να υποστηρίξει την Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε απλώ και μόνο επιμέρου συστήματα που θα βελτιστοποιούν ορισμένε διαδικασίε, αλλά δεν θα αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για αυτέ τι ε, μεγάλε, αν θέλετε, εξελίξει ε, τι οποίε σα ανέφερα. Και αυτό το αναφέρω γιατί συχνά ακούμε εδώ στις Βρυξέλλες ότι ότι δηλαδή το, το, το, το τρένο, αν θέλετε, των δεδομένων, όλη αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε μείνει πίσω. Όχι, τα δεδομένα τα οποία πραγματικά χρειαζόμαστε για την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουμε να τα παράγουμε τώρα. Δηλαδή, το, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των δεδομένων που θα χρειαστούμε για τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη του μελλοντο δεν τα έχουμε ακόμα, δεν παράγονται ακόμα. Άρα λοιπόν, ε, ε, ε, σε ό,τι αφορά τι εφαρμογέ που χρειαζόμαστε, έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικό ε, μειονέκτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώ μπορούμε επιχειρησιακά να αξιοποιήσουμε τα υφιστάμενα συστήματα. Εδώ αναφέρουμε στον κατάλογο αξιολόγηση μα ε, κάποια ζητήματα όπω έχετε εφαρμόσει συγκεκριμένε τεχνικέ οι οποίε θα μείωναν το κίνδυνο, για παράδειγμα, δυσμενών διακρίσεων ή ανισότιμη άδικη εντό εισαγωγικών μεταχείρισης. εδώ θα σας αναφέρω και μια συγκεκριμένη περίπτωση για να είμαι σύντομο. Η Microsoft λοιπόν πριν από ε, κάποιε ε, μήνε διοργάνωσε μια μεγάλη διάσκεψη σε ό,τι αφορά την επιστήμη πληροφοριών, το data science. Και αναφέρθηκε κάτι το οποίο ε, θα σας εκπλήξει εσά και ως μέλη του, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Γιατί αναφέρθηκε ότι πρόσφατα επισκευάσαμε, αν θέλετε, ή φέραμε σε πέραση, καταφέραμε να διευθετήσουμε το ζήτημα του fairness, της δίκαιης μεταχείρισης, της όντιμης μεταχείρισης. Τι σημαίνει όμως αυτό ακριβώς, γιατί βέβαια δεν υπάρχει μια, μια, ένας ενιαίος ορισμός του fairness. Αυτό όμως που προσπαθούμε ε, να κάνουμε και αυτό που μας αφορά εδώ είναι ένα, ένα, αυτό το quantitative fairness metrics. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λέμε στον αλγόριθμο μας ε, τι θα πρέπει να κάνει για να λαμβάνει υπόψη του την ισότιμη μεταχείριση, τι πρέπει να κάνει ε, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη την υπερβολική εκπροσώπηση ορισμένων ομάδων του πληθυσμού και ούτω καθεξής. Δεν εγγυώνται όμως αυτά τα μέτρηξ πράγματι αυτή την αποφυγή των δυσμενών διακρίσεων. Άρα λοιπόν ε, στην νομοθεσία μας, ανάμεσα στο ένα και το άλλο άκρο, θα πρέπει να, να, να, να βρούμε το κατάλληλο μέτρο. Δηλαδή το ένα άκρο είναι να πούμε στι διάφορε επιχειρήσει ότι αν εφαρμόσουν τι διάφορε πρακτικέ σε ό,τι αφορά τη σημερινή μεταχείριση, τότε θα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Θα είναι προστατευμένε αυτέ οι επιχειρήσει. Ε, δηλαδή, κατάλληλη εφαρμογή τη ε, δεοντολογία. Δηλαδή, όταν κανεί σχεδιάζει ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη αυτά τα αισθήματα. Το άλλο άκρο ποιο είναι. Πάντοτε παρέχεται προστασία στον τελικό χρήστη έναντι οποιασδήποτε βλάβης. Ανεξαρτήτως δηλαδή του, της δεοντολογίας την οποία πράγματι τήρησε ή όχι ο, ο, εκείνος που ανέπτυξε το εν λόγω σύστημα. Άρα λοιπόν η πρώτη από αυτές τις προσεγγίσεις θα, ήταν, ε, θα θεωρηθεί πολύ εμ, υποστηρικτική της καινοτομίας, ενώ η δεύτερη θα θεωρηθεί ως υπερβολικά προστατευτική η ε, πλήρω προστατευτική του τελικού χρήστη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Ω προ το τι θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων στο επίπεδο σχεδιασμού του συστημάτων και από την άλλη πλευρά το τι θα πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων σε ό,τι αφορά δηλαδή τυχόν ζημίε που θα επιφέρει ένα τέτοιο αλγόριθμο σε ένα σύστημα. Δηλαδή όσο κι αν, ένα, ε, και, και αν είναι ε, σχεδιασμένο για να είναι δίκαιο ένα τέτοιο σύστημα, μπορεί να είναι άδικο. Για παράδειγμα, υπάρχει το, η περίπτωση των flash ε, crashes, δηλαδή περιπτώσει όπου δύο αλγόριθμοι είναι αντίθετοι μεταξύ του, παρότι ο κάθε ένα ξεχωριστά έχει σχεδιαστεί με τον σωστό τρόπο. Παρόλο αυτό όμω, ε, υπάρχουν, ε, αρχίζουν δηλαδή ο ένας να καταρρύπτουν ο άλλος, να ακυρώνουν τον άλλο και έχουμε για παράδειγμα μείωση του, του δίκτυ κατά πόσες μονάδες μέσα σε 10 λεπτά. Και παρότι υπάρχει τεράστια, τεράστιες απώλειες εδώ, ε, δεν υπάρχει κανένας πραγματικά υπέτειος για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν εδώ ε, ε, οι επιχειρήσει θα πούν ότι εμεί ασχολούμαστε με τι διαδικασίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί με το σύστημα τη διακυβέρνηση, τη γενικώ διακυβέρνηση αυτών των διαδικασιών. Και ε, σε αυτόν τον κατάλογο λοιπόν αξιολόγηση, ο οποίο είναι και δημοσιευμένο, περιλαμβάνουμε μία σειρά από ερωτήματα. Για παράδειγμα, έχετε λάβει υπόψη σα αυτή την πτυχή. Έχετε, για παράδειγμα, δημιουργήσει μία ομάδα καθοδήγηση ακριβώ η οποία έχει και την απαραίτητη εκπροσώπηση από διαφορετικέ ομάδε έχετε δημιουργήσει ε, διαδικασίες οι οποίες ε, ε, αποτρέπουν ακριβώς τέτοιους, τέτοιου διαδικασίες δυσμενών διακρίσεων γιατί κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και παράνομες παρότι δηλαδή ο αλγόριθμος αυτός κάθε αυτός μπορεί να είναι τέλειος εντός εισαγωγικών. Άρα λοιπόν αυτή η λίστα αξιολόγηση που έχουμε δημιουργήσει προσπαθεί έστω πρόχειρα, έστω ως πρώτη φάση να θέσει τις παραμέτρους σε ό,τι αφορά το πώς θα πρέπει να σχεδιάσετε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς, επίσης, ως ομάδα εμπειρογνωμόνων, έχουμε βασιστεί και στις εργασίες μιας υποομάδας ε, σε σχέση με έναν ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δεν περιλαμβάνει μόνο το machine learning. Έχει να κάνει με οποιοδήποτε σύστημα το οποίο είναι σε, ε, σε, σε, να συλλέγει δεδομένα και να βρίσκει τρόπους επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων και να ε, δίνει συστάσεις σε ό,τι αφορά την ανάληψη δράσης. Ε, ε, και μπορώ να σας δώσω λοιπόν το link σε ό,τι αφορά αυτό το έγγραφο που περιλαμβάνει τον ορισμό της τεχνικής νοημοσύνης και δεν ήταν εύκολο να, καταλήξουν σε έναν κοινό ορισμό οι εμπειρογνωμόνες. Τώρα, ε, είπατε σωστά ότι αυτές οι συστάσεις δεν προορίζονταν για την, να χρησιμεύσουν ως βάση για την διατύπωση ε, πρόταση πρότασης κανονισμού. Δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να, να λειτουργήσει ως σύστημα αυτοαξιολόγησης, αλλά έχουμε κατευθυνθεί ε, προς κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι που θα μπορούσε να ε, λειτουργήσει επιχειρησιακά στο πλαίσιο και ακριβώς ενός ε, κανονισμού. Και εγώ, επειδή ακριβώς δραστηριοποιούμε και σε αυτό το τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας, γνωρίζω το πώς κάτι τέτοιο θα πρέπει να διαμορφωθεί για να είναι εφαρμόσιμο στην πράξη, σε επίπεδο νομοθεσία. Ε, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ε, τι προκλήσει εδώ ε, και το έχω αναφέρει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πω είναι δύσκολο αυτό και θα πρέπει να γνωρίζουμε ευθύ εξ αρχή ποια είναι η πρόθεσή τη. Δηλαδή το πώ θα αναθεωρήσουμε εμεί αυτόν τον κατάλογο αξιολόγηση, τη λέξη αξιολόγηση, θα εξαρτηθεί ακριβώ από το, την προβλεπόμενη χρήση, αν θέλετε, αυτή τη λίστα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τώρα του stakeholders και τη διαβούλευση με αυτού, αναφέρθηκε επανειλημμένα ότι αριθμητικά τουλάχιστον πράγματι υπάρχει μεγαλύτερη προσώπηση του, τον, του βιομηχανικού κλάδου σε σύγκριση με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Και αυτό που εγώ μπορώ να σα πω από τη δική μου πλευρά είναι ότι δεν έχω κάποια ατζέντα κρυφή από τη δική μου πλευρά. Θέλω απλώ να κάνω τη δική μου δουλειά. Πράγματι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από πλευρά των επιχειρήσεων και, των, και των πολιτών, αλλά εμεί στην ομάδα εμπειρογνωμών υψηλού επίπεδου έχουμε τι απαραίτητε δικλείδε ασφαλείας. Δεν έχουμε επιτρέψει δηλαδή σε κανένα να επιβληθεί στη συζήτηση. Δεν έχουμε επιτρέψει στι επιχειρήσει να το κάνουν. Ε, και γνωρίζετε ότι το, αυτό έχετε διαπιστώσει ότι μιλάω πολύ, οπότε και σε αυτές τις συζητήσεις ε, πάντοτε ε, όταν άκουγα πολύ μονομερείς τοποθετήσει, εξέφρασα τη δική μου άποψη και προσπαθώ από την δική μου πλευρά να συμβάλλω στο να δημιουργήσουμε κάτι θετικό για την Ευρώπη. Ε, και βέβαια αντιλαμβάνομαι αυτό που θα πείτε, ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε κάτι περισσότερο από την ε, καλή θέληση των συμμετεχόντων. Αυτό που μπορώ όμως εγώ να σας πω είναι ότι δεν μας μεταχειρίζονται, αν θέλετε, ε, κάποιες κρυφές δυνάμεις. Δεν είμαστε μαγιονέτες τους. Δηλαδή προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας και τα όσα μας λέει η κοινωνία των πολιτών, Και θεωρώ πως οι διάφορες ακριβώς οπτικές γωνίες των διαφόρων εκπροσώπων σε αυτή την ομάδα ε, δημιουργούν την καλύτερη, ε, μια καλή ισορροπία. Γιατί πραγματικά θεωρώ πως έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία κατά τη δική μου άποψη ε, μέχρι στιγμής. Και στο πλαίσιο της αναθεώρησης που θα κάνουμε των κατευθυντήριων ε, γραμμών ε, θα ε, λάβουμε υπόψη μας και την ταξινόμηση των κινδύνων, την εράρχηση των κινδύνων που δημοσιεύτηκε από, το, από τη Σχετική Επιτροπή Διοντολογίας της, της Γερμανίας. και εγώ δηλαδή θα κάνω μια προσπάθεια από την δική μου πλευρά. Άλλε τρει ερωτήσει έχουμε, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Ναι, ναι, ναι, τώρα κλείνω, κλείνω. Όσον αφορά αυτού του ηθικού αλγορίθμου και του μη ηθικού αλγορίθμου. Διότι είναι ακόμα πιο σύντομα ένα παράδειγμα τέτοιων αλγορίθμων είναι οι αλγόριθμοι οι οποίοι ενσωματώνουν κάποια δεδομένα για τέλο πάντων έλλειψη αντικειμενικότητα, μεροληψία και μπορεί να σχεδιαστεί ένα τέτοιο που να ενσωματώνει ε, κάποιες προκαταλήψεις κατά τέλο πάντων που οδηγούν σε τιμέ διακρίσει, αυτό τα αξίζουν καθημερινή ζωή και αυτό μπορεί ρητά να περιέχεται στον αλγόριθμο. Έλεγχη για συγκεκριμένε ομάδε, για κάποιε συνήθειε, παραδόσει, για κάποιου που έρχονται από συγκεκριμένε γειτονιέ. Δεν μπορούσαμε να σα πω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Οπότε, ποια δικαιώματα προσβάλλονται, έχουμε κάποιε συστάσει πολιτική και έχουμε επίση και μία σύσταση ότι οι πολίτε ε, πάντοτε θα πρέπει να έχουν μια εναλλακτική για να μπορούν να ε, ποντάρουν στο να έχουν κάποιον συνομιλητή άνθρωπο για να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις όσον αφορά ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μη επιθυμητό επιθυμητό όχι μόνο από τη δική του πλευρά, αλλά γενικά να είναι παραβίαση του δικαιώματο και επίση στοιχείο διακυβέρνηση οποιοδήποτε να πείσει με τη νοημοσύνη θα πρέπει ε, από χέρι να προβλέπει κάποιο είδου ε, ένδικα μέσα σε αυτούς των οποίων θίγεται η καθημερινή ζωή. Έχουμε άλλες τέσσερι ερωτήσει, λέει όμω η πρόεδρο. Σύντομα, σύντομα, αν μπορείτε να τα διατυπώσετε και εσεί μετά επίση, κύριε Ρέντερ, να μα τα πείτε σύντομα. Thank you, uh, να τα πω στα γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδελεχή αυτό που μας εξηγήσατε. Μια παρατήρηση και μια ερώτηση έχω κύριε Ρέντα, και τα είπαν και οι συνάδελφοι κάτι που ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Η παρατήρηση μου είναι η εξή. Με την τεχνητή νοημοσύνη, για πρώτη φορά έχουμε αυτές τις μεγάλες τεχνολογικές ρήξεις και στη βιομηχανία, που είναι κάτι όμως που δεν βρήκε σύμφωνη την πολιτική, γιατί παλιά αυτή η ρήξη οδηγούσε σε θέματα υποδομής και αυτό ήταν επιθυμητό από την πολιτική τάξη. Τώρα όμως να δούμε πώς θα αντισταθμίζεται αυτή η νέα τεχνολογία στη νέα βιομηχανία. Θέλουμε μια νομοθεσία που να μην ξεπερνιέται από τις εξελίξεις και αυτό να αφορά και την ε, πολιτική και έτσι να οδηγούμεθα στην κατάλληλη νομοθεσία. Όπως είπατε, προσπαθούμε προσπαθούμε να, να προλάβουμε εκ των υστέρων με νομοθετικές εξελίξεις τις τεχνολογικές. Να δούμε τη τεχνολογία τι διακυβέματα θέτει. Και υπάρχει και κάτι άλλο συγκεκριμένο που δεν ξέρω αν το είπατε, το θέμα δηλαδή της αναγνώρισης χαρακτηριστικών προσώπου και τα σχετικά ζητήματα. Και αυτό ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ιδιωτικό τομέα, αλλά και από το κράτος και από διάφορους φορείς. Οπότε, είδατε τι γίνεται. Αυτό που γίνεται ας πούμε, στην Κίνα μας προβληματίζουν για αυτή τη νέα τεχνολογία. Χρησιμοποιείται αυτή τη τεχνολογία στο αεροδρόμιο των ΗΠΑ, αλλά θέλει και ο δυτικός τομέας να το χρησιμοποιήσει για τα φυσικά πρόσωπα. Οπότε αναδύονται θέματα και για την ασφάλεια και λοιπά, Για τα φυσικά πρόσωπα. Οπότε για αυτά τα προβλήματα τι θα πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο τι πρέπει να κάνουμε για αυτό το θέμα. Είναι και θέμα της κοινή γνώμης. Φοβάται ο κόσμος. Thank you very much. Um, the next question is from Madam Η επόμενη ερώτηση, λέει ο oh, Ευχαριστώ πολύ για τις ε, απαντήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, κάτι που με έκανε εντύπωση και σε αυτά που είπατε και στις γραπτές απαντήσεις είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και μηχανημάτων. Θέσατε το θέμα της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και αναφερθήκατε στις αξίες που έχουμε εδώ στην Ευρώπη που δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική βάση. Όμως και ο προγραμματισμός ενός μηχανήματος. Η τεχνική βάση λοιπόν χρήση των αλγορίθμων και αυτή πρέπει να βασίζεται σε αυτές τις αξίες γιατί ξέρουμε ότι μετά οι μηχανές κάνουν αυτοπρογραμματισμό που μπορεί να απομακρυνθεί από τις αξίες αυτές. Πόσο θα περιορίσουμε αυτό το ενδεχόμενο και ποιος έχει την ευθύνη για να υπάρχει τελικά διαφάνεια. Ποιος αλληλεπιδράσει τελευταία ανάλυση με ποιον. Πώς ε, λαμβάνουν χώρα αυτές τις διαδικασίες. Ποιοι δημιουργούν το πλαίσιο για αυτές τις αλληλεπιδράσεις και κάτι που είναι η βασική μας αρχή. Η ελευθερία του ενός ε, σταματάει στα όρια του, της ελευθερίας του άλλου. Πώς ε, θα διασφαλίσουμε και πώς θα ελέγξουμε την τήρηση αυτών των ε, θεμελιωδών ελευθεριών. Νομίζω ότι η λέξη εμπιστοσύνη, διαφάνεια και ενημέρωση, ανάγκη ενημέρωση, ποιος και σε τι επίπεδο αλληλεπιδρά με ποιον, είναι τα τρία βασικά θέματα. Και το ερώτημα μου είναι ποιος τα ελέγχει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρέντα για την πολύ σφαιρική ε, εισαγωγή του, η οποία ήταν και μακροσκελής και σύντομη. Γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που συζητάμε. Ε, για να είμαι σύντομο, εγώ θα ξεκινήσω παίρνοντα σαν βάση στο συλλογισμό μου τι εξή αρχέ, α το πούμε. Ότι η πρόοδο γενικά, αλλά και η τεχνολογική και η κοινωνική πρόοδο, είναι μια αντιφατική διαδικασία, προχωρά μέσα από αντιφάσει, όμω πάντα πηγαίνει από ένα χαμηλότερο προ ένα υψηλότερο σημείο, από ένα λιγότερο περίπλοκο σε ένα πιο περίπλοκο ζήτημα. Πρώτο. Δεύτερο, ότι η τεχνολογία, η επιστήμη, τα επιτεύγματά τους, κατά την άποψή μου, πρέπει να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να ελαφρύνεται, και να περιορίζεται και να απαλήφεται ο ανθρώπινος πόνος, το τι υποφέρουν οι άνθρωποι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. Πράγμα το οποίο σε μια καπιταλιστική ελεύθερη αγορά, όπως όλοι μπορούμε να δούμε, δεν συμβαίνει. Ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα αυτών πατενταρίζονται, ε, χρησιμοποιούνται εμπορικά με αποτέλεσμα ε, τα τραγικά στοιχεία που έχουμε πια και με αριθμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρώπη γενικά δεν υπάρχει, υπάρχει η Ευρώπη ειδικά. Ε, και στην παρούσα φάση έχουμε 100 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, αρκετά δεκάδες εκατομμύρια ανέργους, 5 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι άστιγοι κτλ. Προβλήματα που όλα θα μπορούσαν να έχουν λυθεί. Έτσι. Άρα λοιπόν ε, καλά κάνετε και κεντράρετε σε αυτούς τους τομείς και ε, η άποψη δική μας είναι ότι θα επιφέρουν συνολικά αλλαγές σημαντικές οι τεχνολογικές εξελίξεις και στο AI, το Artificial Intelligence, σε όλους τους τομείς. Κυρίως στην βιομηχανία, στην κατασκευή, στις υπηρεσίες και σε άλλους τομείς. Ε, και ήθελα να βάλω ένα ερώτημα πιο συγκεκριμένο. Ε, από νομικής άποψης, επειδή εδώ είναι και αυτή η επιτροπή που είμαστε. Τι εκτιμάτε εσείς σαν ερευνητής του κλάδου ότι θα έπρεπε να γίνει, νομοθεσία που θα έπρεπε να προταθεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κυρίως τα δικαιώματα αυτών που παράγουν σήμερα, των εργαζόμενων δηλαδή της διανοητικής και της χειρονακτικής εργασίας, οι οποίοι θα έρθουν να πληγούν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε ένα πλαίσιο καπιταλιστικής ελεύθερης αγοράς τη στιγμή που βλέπουμε ότι η κατεύθυνση είναι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίρνονται μέτρα τα οποία έρχονται ενάντια στα δικά του συμφέροντα. Διαλύονται οι συλλογικέ συμβάσει εργασία, αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότηση, ολοκληρώνω. Αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότηση αντί να μειώνονται. Και όλα αυτά πρέπει κατά την άποψή μου να τα πάρουμε υπόψη, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να μην γενικεύονται, για παράδειγμα, ε, οι ανάγκε να παίρνουμε μέτρα για να καταπολεμήσουμε την ψηφιοποίηση της οικονομίας η οποία δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους άρα να λυθεί προ όφελο αυτό που λέμε κατά τη δική μα άποψη της εργατικής τάξης και των εργαζομένων σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ. Πόση ώρα διάθεσή μου. Δύο λεφτά, δύο λεφτά, εάν μπορείτε. Καλά, καλά, θα προσπαθήσω να είναι πάρα πολύ σύντομο και θα, θα πρέπει κάτι να τα πούμε, να, να τσιμπήσουμε κάτι και να τα πούμε εδώ στι Βρυξέλλε. Είμαι οπότε μπορούμε να τα πούμε και για την αναγνώριση. Ε, βέβαια, είναι μια τεχνολογία που υφίσταται πολλά, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του κόσμου σε πάρα πολλέ απόψει, αλλά επίση ε, είναι και κάποιο είδου ε, άλμα, διότι όταν κανείς το χρησιμοποιεί για τα δικά του δεδομένα, τότε μπορεί να ελέγξει τι γίνεται, αλλά όταν χρησιμοποιείται γύρω-γύρω, τότε αυτό μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Οπότε, ξέρω πάρα πολύ καλά ε, τα, τα ρίσκα αυτού του τη μαζική εποπτεία παρακολούθηση και γιατί έχω μελετήσει το τι γίνεται στην Κίνα και είναι το σύστημα πάρα πολύ αποτελεσματικό των Κινέζων. Επίσης, πάρα πολλοί από τους δικούς μας ε, νόμους διαπώνται από την αρχή της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε ότι κάποια πράγματα που βελτιώνουν την ε, αποτελεσματικότητα πολλές φορές αντισταθμίζονται από την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι αυτά που τώρα προτείνονται, δηλαδή διαφάνεια και επικοινωνία για την ε, αναγνώριση του προσώπου, όλα αυτά που τώρα θα αρκέσουν ήδη. Έχουμε πάρα πολλούς ε, νόμους που έχουν ε, θεμέλιο την επικοινωνία της πληροφορίας και οι χρήστες είναι πάρα πολύ καλοί στο να τα παρακάμπτουν, τα ας πούμε, τι GDPR, δεν αρκεί το GDPR, γιατί τι, τι έχουμε, έχουμε βλώσει αυτό το παράθυρο σε ένα website που εντάξει καλά όλοι λέμε θέλουμε να συνεχίσουμε, λέμε αποδέχομαι και τελειώνει. Οπότε για να αναγνώριση του προσώπου στα ίδια χναρία πάει. Οπότε εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη μετώση του προβλήματος τότε δεν είναι καλά τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί και άλλος τρόπος αντιμετώπιση προβλήματος. Το θέμα είναι περίπλοκο και νομίζω ότι χρειάζονται ε, περισσότερες δηλές ασφαλείας, ιδίω όσον αφορά αυτό που θέλω να πούμε επαναπατρισμό των δεδομένων για τον τελικό χρήστη, αλλά και άλλες δικλείδες. Το άλλο θέμα αφορούσε τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Ένα και μόνο θα σας πω. Α, και αυτό θα μπορούσε να είναι θέμα διδακτορικού. Η σχέση ανθρώπων μηχανών το έχουμε προσεγγίσει ούτως ώστε να είναι ανθρωποκεντρικό το η αντιμετώπιση ανθρωποκεντρική, γι' αυτό βέβαια φαίνεται στενή αντιμετώπιση, γιατί πολλές φορές είναι το θέμα γαλαξιακού επίπεδου. Και στην ομάδα μας αρνούμεθα τον πειρασμό του να δώσουμε αρμοδιότητες, καθήκοντα, πρωτοβουλίες στις μηχανές. Και εμείς μαθαίνουμε προχωρώντας, δηλαδή το θέλουμε τελικά να μπορέσουμε να υπάρχει ένα εργαλείο, κάτι που να μην έχει πολύ αυτονομία. Και αυτή η μηχανή να σχετίζεται με άλλες μηχανές, αλλά ζητούμε από νομικά και φυσικά πρόσωπα να αναλάβουν τις ευθύνες τους για κάποια απόφαση του να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία που θα οδηγήσει σε τέτοιες εξελίξεις και να συνεχίσουν να προσέχουν, να υποπτεύουν αυτό που κάνανε αυτό που κάνανε τι βγάζει για την κοινωνία. Α, αυτό κάνουμε τώρα. Όχι, δεν έχουμε στοιχεία ότι αυτοί οι αλγόριθμοι που μαθαίνουν μόνοι τους θα φτιάξουν δικούς τους κανόνες. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος που μπορώ να σκεφτώ όταν με ρωτάτε για την καταστροφική συνέπεια της τεχνολογίας είναι να, έτσι στην πλάκα να βάλουμε έναν οικονομολόγο να τα ρυθμίσει Ναι, ναι, ναι, η κοινωνική πρόνοια να αυτοματοποιηθεί. Άλλοι μόνο μας όταν βάλουμε την κομμολογία, γιατί όμως έτσι είναι δυνατόν οι αλγόριθμοι μεταξύ τους. Δεν έχουν δική τους ευφία, αλλά είναι απρόβλεπτοι. Ε, επομένως, αυτό είναι ένα από τα θέματα. Πρέπει να επιλύσουμε την ευθύνη, το πάνω χέρι να το έχουν οι άνθρωποι. Η διακυβέρνηση να είναι με συνεχείς επικαιροποιήσεις. Έτσι θα αντιμετωπίσουν τους ε, κινδύνους. Δεν ξέρω αν θα είναι μια ομάδα, κάποιοι ε, εμπλεκόμενοι, αν θα είναι η υπηρεσία που ζητήσει εδώ και 12 χρόνια. Α, όμως ό,τι θα πρέπει να γίνει και βέβαια υπάρχει εδώ κάποιο ρίσκο από αυτούς που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Το λέμε αυτό επένδυση. Επένδυση πολιτικής. Δεν θέλουμε το θέμα να εκτραπεί από αυτά τα κανάλια. Διακυβέρνηση και να το, περισ... να το θωρακίσουμε έτσι που να μην πάρει ανεπιθύμητες ε, επεκτάσεις. Για τη δική σας ερώτηση κύριε, έχω να σας πω το εξή κύριε Λαβάνο. Αυτό που είπα στην υπόλοιπη ομάδα μας τον Ιούνιο που κάναμε την πρώτη μας συνάντηση. Μας είπανε, έχετε εντολή να μας πείτε πώς θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Τους είπα. και δεν συζητάμε πώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε και το θεματολόγιο του 2030. Για να αναρωτηθείτε, πώ θα εξασφαλίσουμε το να γίνει η Ένωση η πιο ανταγωνιστική για τη ρομποτική όσον αφορά την βιομηχανία. Πώ το ξέρω, βιομηχανικό Ιντερνετ, πώ το λέμε. Τέταρτη γενιά βιομηχανία δηλαδή. Και έτσι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα ρομπότ στα εργοστάσια. Για όμως ε, αναρωτηθείτε Πώς η τεχνητή να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να έχουμε την ε, απασχόληση για όλους. Εμ τελείως άλλη απάντηση θα δοθεί σε αυτό το ερώτημα. Άρα εδώ καλείται το Κοινοβούλιο να συνεχίσει, να συνεχίσει να προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι mainstreaming ε, για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς έχουμε πολιτικές μόνο με ανταγωνιστικότητα και κόστος όφελος. Όλα αυτά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, το περιβάλλον, όλα αυτά να τα λαμβάνουν υπόψη. Πολύ δύσκολο αυτό, τα ξέρουμε. Ε, τέτοια κοινωνία θέλουμε. Τέτοια κοινωνία θέλουμε να έχουμε σε 10 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ την Επιτροπή μας και με βάση αυτά που ακούσαμε θα συνεχίσει να μας ενδιαφέρει. Ίσως λοιπόν να σας ακούσουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ε, μας αφιερώσατε τόσο χρόνο. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα και έχουμε καθυστέρηση, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οπότε να περάσουμε τώρα στο σημείο 8. Για την επικουρικότητα δεν έχουμε τίποτα. Οπότε περνάμε στο 9. Είναι ο Γενικός Προπολογισμός της Ένωσης, ε, δικαστήριο, συζήτηση επί του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Ο κύριος Λεμποετών είναι ο εισηγητή για αυτό το θέμα. Οπότε να σα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από αυτήν την τόσο συναρπαστική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, να επανέλθουμε στα συνήθη θέματά μας. Είναι αυτές οι γνωμοδοτήσεις που κάθε χρόνο χρειάζεται να υποβάλλουμε προ την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού στο αφορά την απαλλαγή για εκτέλεση του προπολογισμού τη Ένωση για το 2018 όσον αφορά το δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω δύο τύπου παρατήρησει Θετικές, γιατί γενικά τα πάει καλά το δικαστήριο, αλλά και κάποια άλλα επί των οποίων έχω περισσότερα ερωτηματικά θετικές ε, εκτιμήσεις, που είναι το μεγαλύτερο τμήμα της γνωμοδότησης, το ποσοστό εκτέλεσης του προπολογισμού είναι πολύ υψηλό. 99,18% πρόοδος ε, σε σχέση με το 98-69% της περσινής χρονιάς. Το ελεκτικό συνέδριο δεν ε, έκανε καμία παρατήρηση για το δικαστήριο. Είναι ένα τη χρονιά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει και αυτό να υπογραμμιστεί. Επίσης, τα δύο δικαστήρια που συναποτελούν το Δικαστήριο της Ένωσης αντιμετώπισαν και έκλεισαν 1.769 υποθέσεις το 2018, αριθμός ρεκόρ. Η δραστηριότητα λοιπόν ε, τα πάει καλά. Και τέλος, η ηλεκτρονική πρόσβαση στο δικαστήριο, το e-Courier, επίσης προχωράει. Όλα αυτά πολύ καλά. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα που δεν είναι τόσο θετικά. Δύο σημεία στη γνωμοδότησή μου είναι τέτοια φύση. Πρώτα απ' όλα το 10, όπου υπενθυμίζουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια είχαμε κάποια ερωτηματικά για την αναγκαιότητα διπλασιασμού του αριθμού των δικαστών. Για τους ε, νέους, αν δεν το γνωρίζετε, έγινε μια πολύ έντονη συζήτηση κατά την προηγούμενη θητεία και ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα ο εισηγητής της Επιτροπής μας που ήταν ένας Πορτογάλος συνάδελφος της ε, ομάδας ε, των ε, φιλελευθέρων είχε οδηγήσει λοιπόν τον εισηγητή να τοποθετηθεί κατά αυτού του διπλασιασμού. Παρ' όλα αυτά υπήρξε διπλασιασμός. Αλλά για να ελέγξουμε ότι όντως χρειάζονταν τόσοι δικαστές σημειώσαμε, όπως γράφει και το Ελεκτικό Συνέδριο στο σημείο 10, ότι μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου του 2020 το Δικαστήριο θα πρέπει να υποβάλει μια έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη λειτουργία του και ιδιαίτερα για την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα αύξησης από 28 σε 56 δικαστές. Αύξηση του αριθμού δηλαδή των δικαστών από 28 σε 56. Να το θυμίσουμε αυτό, να μην ξεχνάμε τι Όντως ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον ως εμπειρία για όσου το θυμούνται πόσο έντονη ήταν αυτή η συζήτηση. Θα το θυμάστε κύριε συνάδελφε. Ούτως ή άλλως, όπως λέει ο συνάδελφος, κάθε εμπειρία είναι πλούτος. Δεύτερο σημείο που δημιουργεί ερωτηματικά το 4. Είναι το σημείο 4. Εδώ είναι λίγο ε, πρόσμενα τα νούμερα. Πόσο ε, κρατάνε οι διαδικασίες. Για το δικαστήριο έχει μειωθεί από 15,7 μήνες έχουν περάσει σε 14,7 αλλά για το πρωτοδικείο αυξήθηκε η διαδικασία. Ήταν 20 μήνες το 18 αντί 16,3 του 2017. Υπάρχει μια βέβαια επίσημη εξήγηση, την υπενθυμίζω. Το 2018 υπήρξαν πολλές υποθέσεις, ε, περίπλοκες. ήταν πιο περίπλοκες οι υποθέσεις που υποβλήθηκαν το 18. Αλλά ήθελα να το επενθυμίσω αυτό. Γιατί είναι το μόνο αριθμητικό στοιχείο που δεν τα πάει καλά. Τώρα κάτι που θα σας πω, δεν θα το γράψω, αλλά θα το πω. Δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι έχει να κάνει με το διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών αυτή η επιμήκυση της ε, διαδικασίας για να κλείσουν οι υποθέσεις. Είναι πολύ νέοι δικαστές και ίσως λοιπόν σε μια πρώτη φάση να ε, επηρέασε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Βλέπουμε πόσο κρατάνε υποθέσεις λοιπόν. Όπως τα καταλάβατε, συνολικά είναι θετικός ο απολογισμός και χρειάστηκε να είμαι κάπως δημιουργικός για να πω κάτι πρωτότυπο, για να πω κάτι ενδιαφέρον ε, που θα απευθύνουμε λοιπόν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, κύριε Λουμπρετό για τι προσπάθειέ σα να είναι ενδιαφέρουσα η γνωμοδότησή σα και για την έκθεσή σα γενικότερα. Έχουμε σχόλια ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τους συναδέλφους. Όχι. Οπότε, προθεσμία για τροπολογίες για την γνωμοδότηση του κ. Λεμπρετών 11 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι. Εάν έχετε σχόλια, προχωράμε σημειώνουμε την γνωμοδότηση αυτή. Το επόμενο θέμα. Το 10. Επικύρωση των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Δικηγική Επιτροπή και την Επιτροπή Προπολογισμών του ΕΟΥΠΟ. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τα ονόματα των εκπροσώπων του Οργανισμού για την Πνευματική Ιδιοκτησία. Σήμερα το πλαίσιο συντονιστές αποφάσισαν να προτείνουν του εξή υποψηφίου για να εγκρίνει η Επιτροπή μα για εκπρόσωπους στο Διοικητικό Συμβούλιο Αλφαβητικά η κυρία Ιζαμπέλ Φελτμάν και η κυρία Μαριέλ Γκάλο και για τον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Προπολογισμού την κυρία Ιζαμπέλ Φέλτμαν, μόνη υποψήφια. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε τώρα επί των υποψηφίων, επί του καθενό. Ηλεκτρονική ψηφοφορία θα χρειαστεί, υποθέτω. Α, ηλεκτρονική ψηφοφορία και για τα δύο αξιώματα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε για την κυρία Ιζαμπέλ Φελτμάν. Κύριε Βός, θέλετε μιλήσετε. Ε, ο κύριος Λεβρετό. Ναι, υπάρχουν δύο ψηφοφορίες. Δεν κατάλαβα. Ξεκινάει η ψηφοφορία, λέει, είπατε ότι έχουμε δύο ψηφίου. Ναι, θα ψηφίσουμε. Και για τις δύο υποψηφίους. Και όποια λάβει τις περισσότερες ψήφους θα είναι τακτικό μέλος και εκείνη που θα λάβει τις λιγότερες ψήφους θα είναι αναπληρωματική. Η Κάρον. Θα ψηφίσουμε για την κάθε μία. Τη μία μετά την άλλη. Ή θα ψηφίσουμε μαζί και θα έχουν η καθεμία άλλο κουμπί δηλαδή στο, στο κουτί μας εδώ το ηλεκτρονικό. Όχι, να με τη σειρά, μία-μία. Λοιπόν, θα πω, κυρία Ιζαμπελ Φέλτμαν, αν θέλετε να ψηφίσετε κυρία Ιζαμπελ Φέλτμαν, θα ψηφίσετε. Συν. Και αν δεν θέλετε να την ψηφίσετε, δεν ψηφίζετε. Και μετά θα πω κυρία Μαριέλ Γκάλο, και αν θέλετε να ψηφίσετε, θα ψηφίσετε συν. Και αν δεν θέλετε να την ψηφίσετε, δεν ψηφίζετε. Εντάξει, δεν ψηφίζουν πραγματικά για κανένα. Για καμία. Εντάξει, ωραία. Παρακαλώ. Αν κάποιο θέλει να συμμετάσχει, αν θέλει να απόσχει, τότε δεν ψηφίζεται καθόλου. Μα δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, ωραία, θα ζητήσω και αποχές ποιοι είναι. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, δεν θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας πριν γίνει η δεύτερη. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για την κυρία Φελτμάν. Αν θέλετε να την ψηφίσετε, παρακαλώ, πατήστε το κουμπί συν. Άρχεται η ψηφοφορία. It does need to be. Sorry, we're waiting for one at the front. Ε, περιμένουμε να ψηφίσει ένας άλλος ακόμη, ένα σημείο. Ωραία. Πέρας. Και τώρα να ψηφίσουμε για την κυρία Μαέλ Γκαλό. Um, and... Ωραία. Πέρας. Και το αποτέλεσμα. I'm afraid we may have to repeat this. Maybe we need... Πώς χρειαστεί να επαναλάβουμε τη αλλά για να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε. Okay, I think this... Λοιπόν, κοιτάξτε δεν ε, πέτυχε η ψηφοφορία. Θα επιχειρήσουμε ένα διαφορετικό σύστημα. Νομίζω ότι το σύστημα ηλεκτρονική ψηφοφορία τη δεύτερη φορά μα έδωσε με αποχέ και άλλα πράγματα. Συγγνώμη που σα μπερδεύω. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε συν για την κυρία Φέλμαν και συν για την κυρία Φέλμαν και μείον για την κυρία Γκάλο. Όποιος θέλει να ψηφίσει για την κυρία Φέλμαν θα ψηφίσει το συν και η κυρία Γκάλο θα ψηφίσει το μείον. Και αν θέλετε να κάνετε αποχή μπορείτε να απόσχετε. Ωραία, λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε 10 ψήφους για την κυρία Φελτμάν, 9 για την κυρία Γκαλό και μία αποχή. Οπότε η κυρία Φέλμαν εκλέγεται ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κυρία Γκαλό ως αναπληρωματικό. Και η κυρία Φέλμαν είναι η μόνη υποψήφια για την Επιτροπή Προπολογισμού. Πρέπει να ψηφίσουμε και για την κυρία ε, Φέλμαν. Ψηφίζουμε λοιπόν γιατί αν θέλουμε η κυρία Φέλμαν να είναι η εκπρόσωπός μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, είναι η μόνη υποψήφια. I think we could have one more vote, but um, I will now. Κοιτάξτε, λείπει μια ψήφος, αλλά θα την κλείσω την ψηφοφορία. 11 είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ως μέλος της Επιτροπής Προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ για την απόφαση αυτή. Ε, είπαμε λοιπόν ότι κλαίγεται η κυρία Φέλτμαν, στους τρεις Περνάμε λοιπόν στο τμήμα τη συνεδρίασή μα που θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Οπότε σα προτείνω να κάνουμε ένα σύντομο πεντάλεπτο διάλειμμα, γιατί κάποιοι θα χρειαστεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Οπότε θα συνεχίσουμε και πάλι τι εργασίε μα στι 5 και 10.